so genau sieht. Ganz so getan. Cominciamo. Ας ξεκινήσουμε. Έχουμε ήδη 10 λεφτά καθυστέρησης. Ήδη μας δημιουργεί πρόβλημα, γιατί πάλι πιεζόμαστε. Με μεγάλη χαρά ε, κυρίσω την έναρξη αυτή τη ακρόαση που την περιμέναμε τόσο για τη συμμετοχή των γυναικών στην τεχνολογία επικοινωνιών και πληροφοριών. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κρόεζα, αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το Γενικό Γραμματέα του ΙΤΟΥ, Μαντούν Τουρέ, που συνεργάστηκαν ενεργά με την Επιτροπή μας για να οργανώσουμε αυτήν εδώ την ακρόαση. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης όλους τους ομιλητές ε, που ήρθαν εδώ σήμερα, καθώς και την κυρία Σάντερ από το Facebook, με την οποία θα συνδεθούμε μέσω βίντεο στις 5 η ώρα το απόγευμα. Η Επιτροπή μας, όπως ξέρετε, συζητάει εδώ και καιρό τους τρόπους για να αυξήσουμε τον αριθμό των εμπειρογνωμόνων γυναικών στον κόσμο των τηλεπικοινωνιών. Το κάνουμε στα πλαίσια της καθημερινής μας δουλειάς, πολιτικό-νομοθετικής, αλλά και με κοινέ πρωτοβουλίες μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επίτροπο ειδικά. Και αυτή τη στιγμή ακόμα κάνουμε σημαντικά πράγματα, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε το εσωτερικό του ορίζοντα 2020. Αυτό θα είναι το πρόγραμμα για την, που είναι το πρόγραμμα για την έρευνα και την κοινοτομία, η ισορροπία των φύλων θα γίνει σεβαστή. Θέλουμε το πρόγραμμα αυτό να συνεισφέρει ούτω ώστε να βρει λύσει για να μειωθεί η ανισορροπία που υπάρχει μεταξύ ερευνητών και ερευνητριών, ούτω ώστε να εκμεταλλευτούμε 100% ε, το ανθρώπινο δυναμικό μα. Σήμερα στην Ευρώπη υπάρχουν 7 εκατομμύρια πολιτών που δουλεύουν στις τηλεπικοινωνίες και περιμένουμε ότι 900 ε, θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν το 2015 στον τομέα αυτό. Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών έχει ένα υψηλό δυναμικό αύξηση σε σχέση με άλλους τομείς ευρωπαϊκής οικονομίας και είναι ένας από τους πιο καινοτόμους και δυναμικούς τομείς. Καθώς και αυτός ο οποίος εστιάζεται περισσότερο στην έρευνα. Στην Επιτροπή ε, Βιομηχανίας και Τηλεπικοινωνιών ε, με αυτή την ευκαιρία ξανατονίζουμε τη σημασία των τηλεπικοινωνιών ε, πέρα από την έρευνα και την καινοτομία και σε αυτόν τον τομέα. Τα επόμενα χρόνια πιστεύουμε ότι θα μειωθεί ο αριθμός των πτυχιών, πτυχιούχων στις, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Και επίσης θα πάρουν σύνταξη πολλοί από τους σημερινούς εργαζόμενους. Χωρίς κατάλληλες πολιτικές, προσαρμοσμένες πολιτικές στην πραγματικότητα ε, της απασχόλησης υπάρχει κίνδυνος ο πιο καινοτόμο και δυναμικός τομέας της Ευρώπης να υποσκαφθεί. Είναι απαραίτητο επομένως να το γνωρίζουμε αυτό και να ενισχύσουμε την εκπαίδευση στην ε, επιστήμη, ε, μαθηματικά, τεχνολογία και να δώσουμε δυνατότητες για καριέρα σε αυτούς τους τομείς και στις γυναίκες. Δηλαδή, περισσότερε γυναίκε θα πρέπει να έχουν κίνητρα για να σπουδάσουν και να δουλέψουν στους τομείς επιστήμης και της τεχνολογίας. Στο γυμνάσιο και το λύκειο, περίπου το 90% των γυναικών ενδιαφέρονται για τις τηλεπικοινωνίες. Παρ' όλα αυτά, αυτό το ενδιαφέρον δεν απεικονίζεται στις ε, επιλογές ε, για σπουδές και δεν επιλέγουν τα κορίτσια αντίστοιχε κατευθύνσει στο πανεπιστήμιο. Επομένω, δεν υπάρχουν αρκετέ γυναίκε που δουλεύουν στι τηλεπικοινωνίε και όπω πάντα συμβαίνει, ελάχιστε ε, βρίσκονται σε υψηλέ θέσει όπου λαμβάνονται και αποφάσει. Ε, δεν θα λύσουμε φυσικά όλα αυτά τα προβλήματα σήμερα, αλλά ε, ελπίζουμε η σημερινή ακρόαση να συνεισφέρει στις ε, Διαδικασίε λήψη των αποφάσεων που είναι εξελίξει και θα μπορέσει να διατηρήσει ζωντανό αυτό το θέμα. Η σημερινή ε, συζήτηση θα δώσει ε, και κίνητρο σε περαιτέρω συζητήσει, για περαιτέρω συζητήσεις, ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τη, τα πρακτικά θέματα, έχουμε δύο μέρη συνεδρίαση. Ε, γυναίκες που η καριέρα τους είναι στις τηλεπικοινωνίες, πώς θα εκμεταλλευτούμε το ταλέντο των γυναικών, και πώς θα βοηθήσουμε τη διαδικασία, πώς θα δημιουργήσουμε δεξιότητες για τις τηλεπικοινωνίες ε, για να αυξήσουμε τη θέση απασχόλησης εδώ. Θα τελειώσουμε 5.30. Επομένως, οι ομιλητές θα πρέπει να σεβαστούν τον χρόνο που θα τους δοθεί. Θα θέλαμε να ακούσουμε επίσης τις απόψεις των διακεκριμένων μιλητών μας και με μεγάλη χαρά θα δώσω το λόγο καταρχήν στο Γενικό Γραμματέα του, της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, τον κύριο Τουρέ, Αμαντού Τουρέ. Ξέρετε, σήμερα είναι η μέρα για τις γυναίκες τηλεπικοινωνίες και είναι μια ε, πρωτοβουλία που την υποστηρίζουν και τα κράτη-μέλη της Ένωσης αυτής της ΙΤΟΥ. Ε, σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ, είσαστε πολύ άριθμοι, που δείχνετε ενδιαφέρον και ελπίζω η συζήτηση αυτή να είναι χρήσιμη και για μας ως θεσμικό όργανο αλλά και για εσάς ως άτομα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Καλό απόγευμα μάλλον κυρίες και κύριοι. Κύριε Σατόρι. Κύριε Μπέρ, Μπάιερ. Κυρίες και κύριοι. Μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά είναι για μένα να είμαι εδώ στις Βρυξέλλες μαζί σας για να γιορτάσουμε την ε, εκδήλωση «Τα κορίτσια στην, ε, στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας 2013. Εδώ στις Βρυξέλλες βρισκόμαστε στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. Γνωρίζουμε όλοι την σημασία και την δύναμη των τεχνολογιών πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών στη ζωή μας. Οι τεχνολογίες ICT παίζουν ένα τεράστιο ρόλο σε όλες τις χώρες μας, είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες, πλούσιες, φτωχές, ανεπτυγμένες και μη. Οι τεχνολογίες ICT είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τις γυναίκες σε όλες τις κοινότητες και ιδίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ακόμα και ένα απλό κινητό τηλέφωνο δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να είναι σε επαφή με την οικογένειά τους και τους φίλους τους. Μπορούν οι γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε κάθε είδους χρήσιμες πληροφορίες και οι τεχνολογίες αυτές μπορεί να είναι και ένα εργαλείο για μάρκετινγκ, για παροχή υπηρεσιών, για εμπορικές υπηρεσίες. Για να κατανοήσετε πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι τεχνολογίες αυτές, μπορούν οι γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε υγειονομικού χαρακτήρα πληροφορίες. Αυτός μπορεί να είναι και ο μηχανισμός που επιτρέπει τις γυναίκες να αντιμετωπίσουν θέματα αναπαραγωγικής υγείας. Χωρίς τις, χωρίς την, τις τεχνολογίες αυτές δεν μπορούν να συζητήσουν τα θέματα αυτά ανοιχτά μέσα στην τοπική τους κοινότητα οι εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μεταδώσουν πληροφορίε στις τοπικές γλώσσες και σε εικόνες ακόμα για να φτάσουμε άτομα τα οποία δεν είναι μορφωμένα ή είναι και αγράμματα. Από την ε, οπτική γωνία της έλξης και όχι της όρθισης πληροφοριών. Τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούν επίσης για να συλλέξουν στοιχεία υγειονομικά, ιδίως σε ό,τι αφορά τα παιδιά, ώστε οι χώρες αυτές μπορούν σιγά σιγά να αναπτύσσουν τις υπηρεσίες τους γιατί δεν μπορεί κανείς να διοργανώσει αυτές οι υγειονομικές ε, υπηρεσίες χωρίς να ξέρει σε ποιους απευθύνονται αυτές οι υπηρεσίες. Οι τεχνολογίες ICT δίνουν επίσης σημαντική δυνατότητα βελτίωσης στην παιδεία από, τα απλά, από τις απλές εφαρμογές που βασίζονται σε μηνύματα που μεταδίδονται στο, με, το τηλέφωνο μέχρι την πρόσβαση σε βιβλιοθήκη σε επιγραμμικού χαρακτήρα. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν σημαντική βελτίωση στον αλφαβητισμό, στην ε, λειτουργία της γεωργίας, τις τεχνικές γεωργίες, στην, τις τεχνικές του επιχειρήν και εφόσον οι περισσότερες γυναίκες στον κόσμο βρίσκονται στο δρόμο, περπατούν το περισσότερο μέρο της μέρας τους, τα κινητά τηλέφωνα τους δίνουν μια τεράστια δυνατότητα να συμμετέχουν στον κόσμο. Η οργάνωσή μου, η Διεθνής ε, Ένωση Τηλεπικοινωνιών, ITU, που είναι ο ειδικευμένος φορέας του ΟΗΕ για τις τεχνολογίες ICT, έχει μια μακρά ε, εταιρική σχέση με την telecenter.org, η οποία είναι μια οργάνωση που θέλει να εκπαιδεύσει εκατομμύρια γυναικών σε βασικές δεξιότητες για τις τεχνολογίες αυτές και εφέτος φτάσαμε σε 680.000 γυναίκες από 147 οργανώσεις που εκπαιδεύονται σε 85 χώρες. Στο περσινό φόρουμ στη Γενέβη είδαμε το βίντεο της Telecenter.org που έδειχνε μια γυναίκα από τις Φιλιππίνες που είχε μεταμορφώσει τη ζωή της. Από το να είναι μια υπηρέτρια στο σπίτι έμαθε να στήσει το δικό της εργαστήριο και τη δική της επιχείρηση ε, γραφίστα. Οι τεχνολογίε ICT είναι και ένα από του καλύτερου μηχανισμού για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των γυναικών και η προστασία του κατά τη βία. Ιδίω τη βία στον οίκο, στο οικιακό περιβάλλον. Κυρίε και κύριοι, σε ένα κόσμο όπου 95% όλων των θέσεων απασχόληση έχουν μια ψηφιακή πτυχή, και όπου υπάρχει <clears throat> μεγάλη και αυξανόμενη έλλειψη δεξιοτήτων στον τομέα ICT, πρέπει όλο και περισσότερες γυναίκες να εμπλακούν στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στη μηχανολογία, στην πληροφορική. Πιο πολλές κοπέλες λοιπόν πρέπει να πάρουν ε, μέρος σε, καρι, σε καριέρες ICT. Θα δημιουργηθούν πάνω από 100, ένα εκατομμύριο θέσεις στον τομέα αυτό στην Ευρώπη, όπως είπε και η πρόεδρο μας το 2013 στον τομέα των τεχνολογιών ICT. Γίνεται κάποια πρόοδος και το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ σήμερα το καταδεικνύει. Είναι ένα θετικό βήμα. Είμαστε όλοι μαζί εδώ σήμερα για να επιτύχουμε τους ίδιους στόχους. Έχουμε όμως πολύ δρόμο να διατρέξουμε. Οι γυναίκες κάνουν τα δύο τρίτα της εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο και πάγουν τα δύο τρίτα ε, της παραγωγής τροφίμων, αλλά παίρνουν μόνο 10% του εισοδήματος σε παγκόσμιο επίπεδο και έχουν μόνο 1% της παγκόσμιας περιουσίας. Το 2013 υπάρχουν πιο πολλές γυναίκες επικεφαλής των εταιριών του Fortune 500 από ό,τι στο παρελθόν. Οι γυναίκες τώρα διευθύνουν πάρα πολλές τεχνολογικού χαρακτήρα εταιρείε όπως είναι η Hewlett Packard, η IBM, η Xerox και η Yahoo. Παραμένουν όμως μόνο σε 21 εταιρείε από τις 500 της Fortune επικεφαλής από τις είναι λοιπόν πολύ μακριά οι γυναίκες από το να επιτύχουν μια μορφή ισότητος. Και αυτό είναι τμήμα της προσπάθειάς μας στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. Το 1932 δημιουργήθηκε ο οργανισμός μας το 1865. Το 1932 είχαμε την πρώτη αντιπροσωπεία γυναικών σε ένα μεγάλο συνέδριο. Το 1965, 100 ε, χρόνια αργότερα, για πρώτη φορά είχαμε μια γυναίκα επικεφαλής αντιπροσωπείας στην ITU. Ακόμα και σήμερα από την πλευρά των κυβερνήσεων υπάρχουν μονάχα 16 γυναίκες υπουργοί από τα 193 κράτη-μέλη της ITU και μόνο 10 από, τα 160, <clears throat> από τις 160 ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο έχουν επικεφαλής τους μια γυναίκα. Παραμένω αισιόδοξο. Είμαι πεπισμένος ότι ακόμα και όπως είναι τα πράγματα, διοργανώσεις όπως η σημερινή όλα αυτά τα γεγονότα που γίνονται σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο και γίνει κάπου 1.500 εκδηλώσεις που γίνονται σε περίπου 100 χώρες. Πέρσι είχαμε 1.200 εκδηλώσεις σε 89 χώρες και έχουμε σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ φέτο, Ακόμα και με αυτό τον αριθμό λοιπόν εκδηλώσεων ελπίζω ότι θα υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια και θα υπάρχουν περισσότερες γυναίκες που μελετούν τεχνολογικά θέματα και θα ακολουθήσουν τεχνολογικές καριέρες. Οι εικόνες από, αυτά τα, από αυτές τις εκδηλώσεις θα δημοσιευθούν στην ε, διαδικτυακή πύλη www.girlsinict.org και με αυτόν τον τρόπο θα παρουσιαστούν πάνω 500 προγράμματα που είναι ε, δίκτυα επιγραμμικά, υποτροφίες, ε, δίκτυα chat και όπου οι γυναίκες μπορούν, ή τα κορίτσια μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα. Μπορώ λοιπόν να σας προσκαλέσω να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα. Από την ε, πλευρά της η Ευρυζωνική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών που δημιουργήθηκε πριν από τρία χρόνια έχει δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας πέρσι το Σεπτέμβριο για την ευρυζωνικές επικοινωνίες και το φύλλο. Μετά από μια έκκληση της ε, Τζίνα Ντέιβις να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε ευρυζωνικέ επικοινωνίες. Ένας από τους κύριους επιτρόπους τη Ευρωπαϊκής Ένωση είναι Νέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα είναι και η επόμενη ομιλήτριά μας. Εμείς χαιρόμαστε που έχουμε ένα τόσο εξέχον, μια τόσο εξέχουσα προσωπικότητα ω μέλος τη ε, ευρυζωνική επιτροπή. Ξέρουμε, μια γυναίκα που τα λέει σταράτα και μας κρατάει στην ζήτα συνέχεια. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρετε εδώ στην Κομισιόν. Το έργο της Ευρωζωνικής Επιτροπής για τις Ευρωζωνικές Επικοινωνίες και το Φύλλο είχε την πρώτη συνεδρία στο Μεξικό πριν από ένα μήνα με επικεφαλής ένα εκπρόσωπο, μία εκπρόσωπο της ε, UNDP και με μεγάλη χαρά ήμουνα και εγώ μέλος, ήμουνα παρόν σε αυτήν την συνεδρίαση με τον Κάρλο Σλιμ και τον πρόεδρο Καγκάμε της Ρουάντα να είναι αντιπρόεδροι αυτής της Επιτροπής. Με τον τρόπο αυτό βλέπουμε ότι υπάρχουν υποδείγματα ρόλων από γυναίκες στον αναπτυσσόμενο κόσμο που έχουν επιτύχει την ισότητα με τους άνδρες. Έχουμε μια κυβέρνηση με 50% άνδρες, 50% γυναίκες Το ίδιο συμβαίνει με το διπλωματικό σώμα, τους πεζευτέ και τα πηγαίνουν πολύ καλά. Για τη Ρουάντα αναφέρομαι. Με το να εργαζόμαστε λοιπόν από κοινού και να χρησιμοποιούμε την κοινή μας θέληση μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο τόπο για να ζούμε και αυτό σημαίνει ότι θα είναι πιο ισοδίκαιος και πιο, ένας πιο πολύ χώρος ισότητος για τις γυναίκες και τα κορίτσια στον τομέα της ICT. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να λάβω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Τουρέ. Είναι Ελικρούς τώρα, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι υπέρ μιας μη ισόρροπης παρακολούθησης των συνεδριάσεων, όχι 50% γυναίκες και 50% άνδρες, αλλά κάτι καλύτερο, αυτό που βλέπω εδώ. Χάρη σε εσά λοιπόν και στην Επιτροπή σας, τα θέματα έχουν αρχίσει και αντιμετωπίζονται σοβαρά. Και αυτό είναι δικαιολογημένο. Όταν έλεγε η μέρνη Μονρό ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος των κοριτσιών. Δεν ισχύει σήμερα μάλλον αυτό. Ο καλύτερος φίλος των κοριτσιών είναι οι ικανότητές τους στον τομέα της πληροφορικής και της τηλεπικοινωνίας. Αν έχετε αυτές τις ικανότητες θα ακολουθούσουν και οι πολύτιμοι λύθοι. Δεν υπάρχει αμφιβολία είναι στο ότι οι εργασίες στον χώρο αυτό ε, αμείβονται με τον ίδιο τρόπο ισότιμα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Θέλουμε περισσότερες γυναίκες λοιπόν εδώ. Έχει μεγάλη σημασία για τις γυναίκες και κάθε γυναίκα θα πρέπει να έχει τα μέσα έτσι ώστε να ελέγχει με τέτοιο τρόπο τη ζωή της σήμερα. Στις τηλεπικοινωνίες οι ικανότητες θα δώσουν νέες ευκαιρίες, καινοτομία και φυσικά παίζει και θετικό ρόλο στην οικονομία μας. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια έλλειψη ενός εκατομμυρίου εργαζομένων βραχυπρόθεσμα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Αυτό τέθηκε και από τον Γενικό Γραμματέα μία από τις ανησυχίες που έχουμε και μία από τις προκλήσεις για το 2015 για την Ευρώπη είναι να προσπαθήσουμε να πληρώσουμε κενές θέσεις με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ικανότητες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Αυτό ισχύει λοιπόν και αν δεν το πετύχουμε μέχρι το 2015 θα χάσουμε πάνω από, μια, από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Αν αποτύχουμε θα βλάψουμε την ανταγωνιστικότητά μας και θα μειώσουμε την απασχόλησή μας. Περισσότερες γυναίκες λοιπόν στον κλάδο αυτό είναι η απόλυτη λύση, αδιαμφισβήτητη λύση. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι εδώ. Το πρόβλημα δεν είναι να πείσουμε τις γυναίκες να χρησιμοποιούν γενικά την πληροφορική και την τεχνολογία. Ε, οι γυναίκες έχουν αρχίσει και το κάνουν αυτό όλο και περισσότερο με ρυθμούς πολύ πιο υψηλούς από τους άνδρες και τις χρησιμοποιούν συνεχώς εντατικά, δημιουργικά και εφάνταστα, περισσότερο εφάνταστα από ότι οι άνδρες, ιδιαίτερα τα κοινωνικά μέσα επικοινωνίες. Από τη Silicon Valley μέχρι τις τενεκεδουπόλεις του Ναϊρόμπι προσπαθούν οι γυναίκες να βελτιώσουν τις δυνατότητές τους και να βελτιώσουν τη ζωή τους, την ίδια τους τη ζωή και τη ζωή των μελών της οικογένειάς τους. Όλοι μας βλέπουμε τις βιομηχανίες να δημιουργούν κάποια προϊόντα ειδικά για τις γυναίκες. Και δυστυχώς πολλές φορές ε, σχεδιάζονται από άνδρες Sometimes the Οι γυναίκες δεν χρειάζονται όμως τέτοιου είδους προϊόντα ειδικά για αυτές. Όπως και δεν χρειάζονται ειδικά αυτοκίνητα ή ειδικά στυλό. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες στις σταδιοδρομίες ε, στο χώρο αυτό λιγότερο από τον ένα στους τρεις εργαζομένους είναι οι γυναίκες. Και αυτό μάλιστα κυρίως σε χαμηλά αμοιβόμενε θέσεις. Χτες παρουσίασα την πρώτη πρωτοποριακή ε, ευρωπαϊκή προσπάθεια βράβευσης των γυναικών επιχειρηματιών στον τομέα αυτό, στον κλάδο αυτό. Πραγματικά εξαιρετικά, ε, εξαιρετική ευκαιρία και ήταν τιμή για μένα που μπόρεσα να δώσω τα βραβεία αλλά και οι 15 πρώτοι ήταν επιχειρηματίες άνδρες. Ε, και αυτό δείχνει φυσικά ότι οι γυναίκες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν, να αλλάξει η κατάσταση. Πολλές γυναίκες κάνουν τεράστιες προσπάθειες ε, για να αλλάξουν τα πράγματα. Να δούμε λοιπόν τι υπάρχει και τι πρέπει να αλλάξει και ευχαριστώ και τις γυναίκες που πήραν μέρος στην προσπάθεια αυτή και θα αναφερθώ σε κάποιες από τις ιδέες που έκαναν προτάσεις. Πολλές φορές θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα σχολεία, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Χρειάζονται τα κομπιούτερς ή υπολογιστές από την αρχή της σχολικής εκπαίδευσης. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους δάσκαλους, πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους καθηγητές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι υπολογιστές σε όλες τις δραστηριότητες. Αλλά το θέμα δεν είναι να αποκτήσει κανείς κάποιες ικανότητες, το θέμα είναι να τις χρησιμοποιήσει σωστά. Και γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν πολλές γυναίκες που έχουν επιτυχία στον τομέα της πληροφορικής και δεν εργάζονται, δεν φεύγουν από την οικογένειά τους. Έστω και λίγες από αυτές τις γυναίκες να γυρίσουν στην εργασία θα δώσουν μια όθηση στην οικογένειά μας, θα είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό θα προσφέρει 9 δις κατέτος σε ετήσια λοιπόν βάση. Χάνουμε λοιπόν σε ετήσια βάση 9 δις κατέτος. Αρκετά χρήματα για να καλύψει κανείς τα επόμενα δύο χρόνια το έλλειμμα. Είναι σαφές λοιπόν ότι απαιτούνται πρότυπα να υπάρχουν συναντήσεις με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με ε, ικανότητες και με σταδιοδρομίες στον τομέα της πληροφορικής. Και είναι πολύ καλό να ξεκαθαρίσουμε ότι η Επιτροπή σας προεδρεύεται από γυναίκα, έτσι δεν είναι. Υπάρχουν γυναίκες ικανές εδώ, υπάρχουν ιστορίες επιτυχίας και κάποιες από αυτές θα τις ακούσουμε αργότερα. Αλλά καλό θα είναι να έχουμε και περισσότερες νέες γυναίκες που συμμετέχουν στην προσπάθεια. Είναι καλό να υπάρχουν πρότυπα και στην, όχι μόνο στον πραγματικό κόσμο αλλά και ε, στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, να υπάρχουν προσδοκίες για τις νέες γυναίκες και να μην μείνουμε στις νεράιδες και στις πριγκίπισσες. Υπάρχουν λοιπόν στη βάση των πραγμάτων πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Η Λίντα Λούκας, η ψηφιακή πρωταθλήτρια της ε, Φιλανδίας, είχε σημειώσει πολύ μεγάλες επιτυχίες και στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, ο Gates έχει ξεκινήσει μια ιστοσελίδα για να συμμετέχουν περισσότερα γυναίκες. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες, να στρέψουμε την προσοχή των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο. Έτσι λοιπόν ο πολλαπλασιασμός αυτών των πρωτοβουλειών στην βάση θα βοηθήσει πολύ. Η πρόθεση πρωτοβουλειών όπως τα ψηφιακά νέα το δίκτυο επιτάχυνσης των, ε, της γυναικείας παρουσίας ε, και διεύρυνσης της γυναικείας παρουσίας στον επιχειρηματικό κόσμο. Οι πρωτοβουλίες για τη γυναίκα στην επιχείρηση. Όλες αυτές θα βοηθήσουν την Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική. Αλλά ας μην σταθούμε πατερναλιστικά απέναντι στο θέμα. Ας προσπαθήσουμε όμως να προωθήσουμε την υπόθεση αυτή δεν είναι οι γυναίκες θύματα που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Έχουν ικανότητες, έχουν ταλέντο και οι οικονομίες μας τις χρειάζεται. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τις γυναίκες αυτές. Δεν μπορούμε εμείς να αφήσουμε να χαθεί το 50% των δυνατοτήτων μας. Δεν είναι θύματα οι γυναίκες, ας συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό, ας το ξεκαθαρίσουμε. Και έτσι θα έχουμε κάνει το πρώτο βήμα για να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα προβλήματα. Όχι βέβαια αγνοώντας την πραγματική φύση της συγκεκριμένης δραστηριότητας του τομέα της τηλεπικοινωνίας και της πληροφορικής, αλλά έχουμε τις ικανότητες, έχετε τις ικανότητες και πρέπει να τις χρησιμοποιήσετε. Ούτε ε, το θέμα είναι να προσελκύσουμε τις έξυπνες γυναίκες ε, ε, ειδικά, όχι το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στη σχέση των γυναικών με την πληροφορική. Υπάρχει όμως μια ευκαιρία, υπάρχει μια δυνατότητα και πρέπει αυτή τη δυνατότητα να την ενδυναμώσουμε, να την μεγενθύνουμε, να βοηθήσουμε τις γυναίκες να ολοκληρώσουν τις προσδοκίες τους. Οι γυναίκες στον χώρο αυτό λέγουν ότι οι, τους, οι σταδιοδρομίες τους είναι ιδιαιτέρως ε, ενδιαφέρουσες, είναι προκλητικές και είναι γεμάτες από ευκαιρίες. Οι γυναίκες μπορεί στον χώρο αυτό να κερδίσουν 9% πάνω από τον διαφορά που έχουν οι αμοιβέ ανδρών γυναικών σε άλλους τομείς. Δεν υπάρχει λοιπόν καλύτερο μέσο για να αλλάξουν τα πράγματα γιατί να προσπαθήσουμε να το αγνοήσουμε αυτό, δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Ας δείξουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Αυτό δεν είναι φιλανθρωπία. Αυτό είναι οι επιχειρήσεις, είναι πολιτική, είναι οικονομική λογική. Οι επιχειρήσεις αυτές που ανήκουν σε γυναίκες, που τις διευθύνουν γυναίκες, έχουν υψηλά εισοδήματα και υψηλές δυνατότητες επιτυχίας και να μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες είναι επίσης και ένα μεγάλο τμήμα της βάσης των πελατών ε, της πληροφορικής αυτής και της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Πρέπει λοιπόν να καλύψουμε το κενό αυτό των γνώσεων στον τομέα σε συνεργασία με τη βιομηχανία, σε συνεργασία με τους παροχείς υπηρεσιών και έτσι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε να αφιερωθούμε στο να αποκτήσουν οι γυναίκες περισσότερες ικανότητες, περισσότερες γνώσεις και να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στις γυναίκες ακόμα περισσότερο. Λίγες περισσότερες ιδέες λοιπόν. Μήπως θα πρέπει και οι άνδρες να εορτάζουν για την παρουσία των ανδρών και των γυναικών στον συγκεκριμένο χώρο ή μήπως να υπάρχει ένα σύστημα καθοδήγησης, ένα δίκτυο καθοδήγησης των γυναικών με τις γυναίκες που βρίσκονται ήδη στο εσωτερικό αυτού του δικτύου και εγώ θα είμαι πρώτη εκεί. Ή ένα νέο πρόβλημα, πρόγραμμα συγγνώμη, επιτάχυνσης της συμμετοχής των γυναικών στον επιχειρηματικό κόσμο. Δεν είναι εύκολα όλα τα πράγματα. Δεν είμαστε μια ομοιογενής ομάδα οι γυναίκες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το να προσπαθήσει κανείς να πλησιάσει τις γυναίκες προαπαιτεί μια ολόκληρη σειρά από μέσα έτσι ώστε να σεβαστούμε τις διαφοροποιήσεις και τις αλλαγές που υπάρχουν σε επίπεδο πολιτικό, σε επίπεδο προτύπων, σε επίπεδο διοίκησης επιχειρήσεων. Ελπίζω τα μηνύματα να μπορέσουμε να τα περάσουμε σε όλες τις γυναίκες και να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Ελπίζω και τα μέλη του Κοινοβουλίου να αναφερθούν στις πρωτοβουλίες αυτές τις εκλογικές τους περιφέρειες. Όπως είπα είναι μια μεγάλη ευκαιρία και εμείς δεν κάνουμε καμιά ιδιαίτερη χάρη στις γυναίκες. Όχι, η βιομηχανία χρειάζεται το ταλέντο των γυναικών. Η οικονομία μας χρειάζεται τις γυναίκες και την καινοτομία τους. Οι ψηφιακές γυναίκες αξίζουν πάνω και πολύ περισσότερο από τα διαμάντια. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε την Επίτροπο Κρούζ και τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, τον Αμαντού Τουρέ, για τις ομιλίες τους και για την παρουσία τους. Και τώρα θα ξεκινήσει το πρώτο πάνελ ομιλητών. Γυναίκες της... στην τεχνολογία πληροφοριών πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το γυναικείο ταλέντο. Η Τζάνα Μαρτινέγκο, η Σάσκια Βαν Ούφελεν και η Μονίκ Μογό θα ήθελαν να έρθουν στο βήμα. Ε, ε, Buongiorno.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 Ideal KTS. Ideal KTS. the Passiamo al nostro... Πολύ ωραία. Ας περάσουμε στο πρώτο πάνελ. Ας δώσω το λόγο στην Τζάνα Μαρτινέγκο, που είναι πρόεδρος της και της οργάνωσης Γυναίκες Τεχνολογία. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Ε, με τιμά πολύ η πρόσκληση αυτή. Ε, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε δημόσια ακρόαση. Είχα την τύχη να δουλέψω πολύ νωρίς ε, για το διάλογο μεταξύ ατόμων και πώς διευκολύνεται από την τεχνολογία. Αυτό το 1983 ε, και ήταν στην καρδιά αυτού που κάναμε στα εργαστήρια τότε. Ε, και σήμερα βρίσκεται στην καρδιά κάθε ανθρώπινη δραστηριότητας. Η πολυάριθμη οικογένειά μου με έμαθε να μπορώ να συμφιλιώνομαι. Ε, η ζωή μου ήταν πολύ επιτυχή χάρη στις τεχνολογίες πληροφοριών. Εγώ από τη φύση μου είμαι αισιόδοξη και κοιτώντας το μέλλον πάντα λέω ότι πρέπει να ανακαλύπτουμε, να μοιραζόμαστε και να ενισχύουμε. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες από μόνες τους μπορούν να δημιουργήσουν έξυπνες πόλεις. Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό ε, με, μια, με ένα βαθύ προβληματισμό της οργάνωσης ε, της κοινωνίας, για μια κοινωνία που, θα, που ούτως ή άλλως αλλάζει με ένα απίστευτα γρήγορο ρυθμό ε, που δεν έχει, τον έχει ζήσει ποτέ η ανθρωπότητα. Ε, με συμμετοχή, η συμμετοχή σε αυτή την ανάπτυξη, η ευέλικτη εργασία, η συνεχής ε, εκπαίδευση, κατάρτιση, η κινητικότητα είναι λέξεις οι οποίες με συνόδευσαν αυτά τα τελευταία χρόνια ως ε, ερευνήτρια και επιχειρηματία. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις λέξεις να δώσουμε ιδιαίτερη αξία που συχνά αλλάζουν ανάλογα με το διαφορετικό πλαίσιο με στο οποίο χρησιμοποιούνται. Και μερικές φορές ε, στις, στις λέξεις αυτές δεν, ε, αυτές δεν τις συνοδεύουμε από νέα μοντέλα ενημέρωσης, πληροφοριών κτλ. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Ετοιμάζουμε φοιτητές για τεχνολογίες και επαγγέλματα που δεν υπάρχουν ακόμα. Και σκεφτείτε, τα πιο σημαντικά επαγγέλματα το 2010, δηλαδή αυτά που τα ζητάει πιο πολύ η αγορά, δεν υπήρχαν το 2004. Μία έρευνα που ζήτησε η Βρετανική κυβέρνηση εντόπισε 20 επαγγέλματα το 2030 και όλα αυτά θα βασίζονται στις τηλεπικοινωνίες. Ε, και ζήτησα εγώ στα, ε, ζήτησα από τα εγγονάκια μου ε, τρία αγόρια, τρία κορίτσια να μου πούν τη γνώμη τους. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη συνέχεια της διηγήσής μου, που όλο, όλη αυτή η διήγηση συγκεντρώνεται. Όλη αυτή η, η ομιλία μου είναι στραμμένη προς το μέλλον, που πιστεύω ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψουμε το μέλλον είναι να το εφεύρουμε. Και νομίζω ότι οι γυναίκε είναι πολύ ευρηματικά και όντα και μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτό. Η ποιότητα τη ζωή ε, το 2030, χάρη σε όσα θα έχουμε κάνει και τι προηγούμενε δεκαετίε, θα είναι καλύτερη μόνο αν οι χώρε έχουν κάνει επιλογέ και συνεχεία πολιτικέ με σκοπό να προωθήσουν την πραγματική καινοτομία, τεχνολογική και κοινωνική, στι επιχειρήσει και στα θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να βελτιώσουν και να υποστηρίξουν την ε, ε, έρευνα και να βελτιώσει το ανθρώπινο ε, δυναμικό. Το λέμε χρόνια αυτό. Τώρα πρέπει να το κάνουμε όμω. Τι πρέπει να κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε και να συνοδεύσουμε αυτή τη ε, διαδικασία τη της ε, ψηφιακής μας αυτής πορεία, πορείας. Σήμερα. Ποτέ όπως σήμερα, σε μια, ποτέ δεν ζήσαμε όπως ζούμε σήμερα σε, σε μια κοινωνία τόσο πολύ ποικίλη, με πολλές γλώσσες κτλ. και πολλές δεξιότητες. Ε, αν τις έχουμε αυτές, κάθε πολίτης μπορεί να είναι πραγματικός πολίτης, να αναπτύξει τις ικανότητες του, να ζήσει αξιοπρεπώς, να εργαστεί αξιοπρεπώς, να συμμετάσχει στην ανάπτυξη της πόλης, του χωριού του, να βελτιώσει τη ζωή του και των άλλων, να πάρει αποφάσεις ε, με τα λόγου γνώσεως και να συνεχίσει να τις να παίρνει τέτοιου τύπου αποφάσεις. Η ψηφιακή ατζέντα, το ψηφιακό θεματολόγιο, χάρη στη δουλειά που έγινε αυτά τα τελευταία χρόνια, μας επιτρέπει να θέσουμε κάποιους πυλώνες που εγώ, με τους οποίους εγώ ασχολήθηκα εδώ και 30 χρόνια. Ε, η πρόσβαση στο ίντερνετ είναι βασικό το δικαίωμα των ατόμων. Ε, η ρύθμιση της εργασίας online. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα ε, τα οποία εγώ τα έζησα ως ερευνήτρια και επιχειρηματία. Συμμετείχα επίσης και ενεργά σε προγράμματα στη δεκαετία του 90, ΕΣΠΡΙ και ΔΕΛΤΑ και είχα τι τώρα ας πούμε το 96 να ξεκινήσω ένα πρόγραμμα ψηφιακή ένταξης για τους λιγότερο ευνοημένους πληθυσμού ε, στη χώρα μου, την Ιταλία. Χάρη στην τεχνολογία σήμερα, οι πόλεις γίνονται όλο και πιο πολύ η καρδιά μια νέας οικονομίας, η οικονομία των υπηρεσιών. Στην Ιταλία το 70% του ΑΕΠ ε, προκύπτει από τις υπηρεσίες. Τα επαγγέλματα τα οποία, τα οποία γενικά χρειάζονται σημαντικές αλλαγές ε, και σε γνώσεις Ούτω ή άλλω έχει γίνει μια μεγάλη αλλαγή τα τελευταία 30 χρόνια και η αλλαγή αυτή αφορά την ε, ένταξη των φυσικών επιστημών, των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και των ανθρωπιστικών επιστημών στις γνώσεις μας και η διασύνδεσή τους. Ε, με αυτόν τον τρόπο στο μέλλον θα έχουμε ε, όλο και περισσότερες γνώσεις από όλο και περισσότερους τομείς. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα που το καταφέρουμε χάρη στην τεχνολογία της πληροφορικής. Συνεχίζουμε αυτή την μικρή διήγηση, προχωράμε, βλέπουμε τα, οι αυτές οι οριζόντιες ας πούμε, για να τις πούμε έτσι, υπάρχουν κυρίως στις γυναίκες. Υπάρχουν ε, γνώσεις που μου θυμίζουν πραγματικά τις γυναίκες, ε, την ε, θέλησή τους να μάθουν. Μερικές φορές είναι και το Παραδείγματο χάρη το ταλέντο της διαμεσολάβησης. Το είδα στη γιαγιά μου και στη μάνα μου. Οι γυναίκες τα, τα κατάφερναν, ειδικά σε αυτούς τους τομείς. και σήμερα η διαμεσολάβηση, όταν έχουμε τόσο περίπλοκα προβλήματα, αυτή η τέχνη της ανεσολάβησης ε, μαζί με άλλες τέχνες έτσι, έμφυτες που έχουν οι γυναίκες είναι φοβερό εργαλείο για να προστατεύσουμε ας πούμε τις μειονότητες, να προστατεύσουμε τις αξίες, τα άτομα, τα δικαιώματά τους. Προχωράμε. Πρέπει να σας πω ότι το πάθος και η συμπόνια είναι έμφυτο στις γυναίκες. Ε, λίγο, οι άντρε δεν τα πάνε τόσο καλά, ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι γενετικό το πρόβλημα. Μείνετε εδώ σας παρακαλώ στην ίδια διαφάνεια. Όλες ε, οι λέξεις στα αγγλικά που ξεκινάνε με το E, δηλαδή electronic, δεν είναι η αλλαγή απλώς μίας λέξης. Δεν αλλάξαμε το tele και βάλαμε το E. Telework, το, να το κάνουμε e-work. Δεν πρόκειται για μια τέτοια απλή ε, αλλαγή λέξης. Πίσω από όλα αυτά τα ε, τα ε, τα αγγλικά, υπάρχει μια τρομακτική αλλαγή, μια ανατροπή που αφορά τις προσωπικές, ανθρώπινες α, γνώσεις και δεξιότητες και τη φοβερή εξέλιξη των τεχνολογιών, ε, τις οποίες παρατηρούμε και βλέπουμε ότι αναπτύσσονται εκθετικά. Η άποψή μου είναι ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών μπορούν να μας δάξουν και άλλα πράγματα. Ε, καινοτομία, όχι μόνο τεχνολογική αλλά και κοινωνική. Και για μένα αυτό το πράγμα είναι σημαντικό. Πιστεύω ότι σήμερα όλο και περισσότερο οι νέες διαδικασίες που βασίζονται στις ε, υπηρεσίες ζητούν, ενέχουν την ανάγκη της επικοινωνίας ε, τεχνολογιών και προσώπων, επικοινωνίας, το τονίζω, το υπογραμμίζω. Διάδραση, διάλογος δηλαδή, συζήτηση, φήμη και συμμετοχή. Δεχτείτε αυτή την, αυτόν τον ολιστικό έτσι, ορισμό της τεχνολογίας των πληροφοριών. Υπάρχουν και μια άλλη σειρά, ε, υπάρχει και μια άλλη σειρά λέξεων που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εδώ έχουμε ένα ε, πρόθεμα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ γνωστές λέξεις τους πληροφορικάριους και που είναι πολύ σημαντικές γιατί ε, πολύ σημαντικές και δύσκολες ε, διαδικασίες ε, λήψης των αποφάσεων, παραδείγματος χάρη οικοδόμηση των έξυπνων πόλεων, είναι απαραίτητες για να ικανοποιήσουν ε, κοινωνικές ανάγκες και εκεί ο καθένας μπορεί να παίξει το ρόλο του. Κλείνω, κλείνω. Ε, γυναίκες εδώ σε αυτή τη διήγησή μα, είναι όπως ο Λεωνάρντο. Έχουμε φτάσει όμως το 2030 και θα σα πω κάτι καινούριο. Ξέρετε ότι ε, γυναίκες και τεχνολογία είναι ένα δίπολο που μπορεί να κερδίσει. Ε, η Νέλη Κρούς έχει δίκιο που λέει ότι είναι ένας πόρος, ένας πλούτος ε, με τεράστιο δυναμικό, όπως και οι νέοι. Και θα πρέπει οι επιχειρήσεις, οι αρχές ε, να τις αξιοποιήσουν. Γιατί είναι στο κέντρο της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής αξίας. Όχι μόνο ότι είναι δηλαδή δίκαιο οι γυναίκες να συμμετέχουν, αλλά είναι και χρήσιμο. Κλείνοντας, θέλω να πω, οι γυναίκες δεν έχουν πετύχει ακόμα την ισότητα. Οι, οι κοινωνίες χρειάζονται α, την πολυμορφία και το ταλέντο. Σας ευχαριστώ πολύ και ε, ζητώ συγγνώμη αν μίλησα πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μαρτινέγκο. Θα δώσω το λόγο τώρα στη Σάσια Βανχούφελαντ. Um, Ευχαριστώ. Καταρχήν ζητώ συγγνώμη δεν ε, σας κουνάω το δάχτυλο, απλώς είναι το σύστημα για να αλλάζουμε διαφάνειες και γι' αυτό δίνω μηνύματα με το δάχτυλό μου. Και μάλλον είμαι η μόνη εκπρόσωπος του ιδιωτικού τομέα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι άμεση σε αυτά που λέω, όπως το κάνω πάντα κάτι το οποίο μπορείτε να αναγνωρίσετε τον εαυτό σας, δεν είναι προσωπικού χαρακτήρα, δεν είναι ηθελημένο. Ο, ο, ο τίτλος του ομιλίας μου είναι πώς να χρησιμοποιήσει κανείς τα γυναικεία ταλέντα. Εμείς ακούμε μόνο αρνητικά πράγματα για τις γυναίκες. Όλα πάνε στραβά, η οικονομία πάει στραβά, όλα δυσκολεύουν, ο κόσμος κουράζεται. Και νομίζω ότι τουλάχιστον η ψηφιακή ατζέντα που προέρχεται από μια γυναίκα επίτροπο είναι θετική. Δεν είναι γκρίνια ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Είναι μια θετική προσπάθεια για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να επιτύχουμε την αλλαγή. Και είναι μεγάλη μου τιμή που θεωρήθηκα η ψηφιακή πρωτοπόρος του Βελγίου και εγώ θέλω να εστιάσω σε τρία σημεία σε όλη την ψηφιακή ατζέντα. Καταρχήν η ψηφιακή ατζέντα στα σχολεία και όχι μόνο στα σχολεία, θα προχωρήσω λίγο περισσότερο γιατί ζούμε σε μια κοινωνία πληροφορίας. Ελπίζω του χρόνου θα έχουμε περισσότερες γυναίκες στην, ε, στις τεχνολογίες ICT και στις ψηφιακές τεχνολογίες. Καταρχήν να προχωρήσουμε σε μια περισσότερη ψηφιοποίηση των σχολείων, Δεύτερον, στο ψηφιακό εμπόριο, αυτό δεν είναι μόνο να πουλάμε παπούτσια στο ίντερνετ. Και τρίτον, να δώσουμε έμφαση στις ε, ηλεκτρονικές δεξιότητες. Γιατί χωρίς αυτές κινδυνεύει κανείς να βρεθεί πίσω από ένα μεγάλο χάσμα. Οι φτωχοί είναι αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Αν δεν δράσουμε σήμερα θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα γιατί θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι προσαρμοσμένοι στην ψηφιακή κοινωνία και απόκληρους ψηφιακά στις κοινωνίες μας. Και αυτό θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Αυτό δεν είναι ίσως η καλύτερη λύση το να κρύψουμε το κεφάλι μας στην άμμο ή αλλιώς μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο και να αρχίσουμε να συζητάμε το θέμα αυτό. Νομίζω ότι η σημερινή πρωτοβουλία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα της ιδέας ότι με την επανάληψη πετυχαίνουμε την τελειότητα. Ότι αν το πούμε αρκετές φορές κάποιοι θα αρχίσουν να κατανοούν ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε κάτι. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Πρέπει να ξεκινήσουμε πάρα πολύ μικροί. Όλοι ξέρουν το παράδειγμα ενός παιδιού δύο ετών που ακουμπάει με τα δάχτυλα του την τηλεόραση και λέει «Μπαμπά γιατί δεν κουνιέται η εικόνα». Πρέπει λοιπόν να θυμηθούμε τον Μεσαίωνα. Τότε μόνο από τα βιβλία μπορούσε κανείς να έχει πληροφορία. Και ο κόσμος της ε, τεχνολογίας επικοινωνιών μπορεί να φαίνεται σε πολλούς παράξενους, είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι συγκεκριμένος για πολλούς και δεν είναι και ιδιαίτερα μοδάτος. Πώς θέλετε λοιπόν οι γυναίκες να μπουν σε αυτό το τομέα αν ήδη στο σχολείο, στο σχολείο τις διδάσκουμε να μην αγγίζουν πράγματα που δεν καταλαβαίνουν. Τι θα κάνουμε λοιπόν με τις νέες κοπέλες. Έχουν μεγάλη ε, ικανότητα καινοτομία και δημιουργικότητα. Μπορούμε να κάνουμε 50 πράγματα συγχρόνως, ακούμε διαφορετικά, δρούμε διαφορετικά. Πώς μπορούμε να τις φέρουμε πιο κοντά στον κόσμο της κοινωνίας των πληροφοριών. Αν θέλετε λοιπόν να προσελκύσετε τις γυναίκες σε αυτό το τομέα, θα πρέπει από <clears throat> μικρή ηλικία να τους εξηγήσουμε ότι αν θέλετε επιτυχία στον επαγγελματικό σας τομέα, αν θέλετε να έχετε επιτυχία σε τομείς που έχουν να κάνουν με ανθρώπινη επαφή όπως είναι ο υγειονομικός τομέας, να αναπτύξετε νέα υποδείγματα στο σχολείο, αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το κάνετε. Μπορείτε να είστε τμήμα αυτού του κόσμου με την προϋπόθεση ότι η οι μελέτες που θα κάνετε, οι σπουδές σας, δεν είναι μονάχα να διαβάσετε βιβλία, παραδείγματος χάρη για να μάθετε αρχιτεκτονική, αλλά να ξέρετε ότι πρέπει να κάνετε σχεδιασμό με υπολογιστή σε τρεις διαστάσεις για να φτιάξετε το μέλλον. Αν το εξη... εξηγήσετε αυτό στα νεαρά κορίτσια, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί για τις κοπέλες το να βοηθούν τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τότε όλα αυτά δεν γίνονται πια βαρετά. Δεν είναι μονάχα για τους ε, μουλούς τους ψωνισμένους της πληροφορικής, αλλά καταλαβαίνουν οι γυναίκες ότι μπορούν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν πράγματα που θα τους οδηγήσουν πράγματι στα διαμάντια, όπως ε, είπε προηγουμένως η ομιλήτρια. Νομίζω λοιπόν ότι με τον τρόπο αυτό, με το παράδειγμα, μπορούμε μπορούμε να προσαρμοστούμε στις δύσκολες καταστάσεις που διατρέχουμε τώρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αν αντιμετωπίσουμε τον κόσμο της αύριο με τους κανόνες του παρελθόν, <clears throat> τότε έχουμε χάσει το τρένο. Το τρένο έχει ήδη φύγει από το σταθμό και έχει εξαφανιστεί. Μπορούμε λοιπόν να φτιάξουμε τις γέφυρες. Μπορούμε να βρούμε τις λύσεις. μπορούμε να είμαστε πραγματιστικές και να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα όχι σε στρατοσφαιρικό επίπεδο, στα σύννεφα, αλλά σε πραγματιστικό επίπεδο. Να δρούμε με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες. Αν θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε την οικονομία πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές, να υπάρξουν οι δεξιότητες των ε, κοριτσιών, και οι άνδρες ακόμα έχουν αυτές τις ε, ικανότητες αν θέλουν να τις εκμεταλλευτούν και αν το κάνουμε αυτό μπορούμε πράγματι να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα που έχουμε σήμερα. Αυτό το οποίο θέλω να κάνω λοιπόν είναι μια ευαισθητοποίηση ως πρωταθλήτρια στα θέματα πληροφορικής. Το λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω και θα το ξαναλέω. Αυτό το ρόλο τον έχω αναλάβει αυτό το Δεκέμβριο. Ένιωσα λοιπόν μεγάλη έκπληξη για το γεγονός ότι οι περισσότερες πληροφορίες που υπάρχουν σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ο γιος μου μιλάει. Είχε πρόβλημα με τα γερμανικά και είναι 15 χρονών και παίρνει τώρα μαθήματα μέσα από το Skype βοήθεια από μια Γερμανίδα καθηγητή. Αυτό είναι ένα είδος ηλεκτρονικού εμπορίου δεν είναι πώληση παπουτσιών, είναι μια ψηφιακή υπηρεσία. Γιατί ο γιος μου είναι, και ο γιος μου είναι πολύ ικανοποιημένο και αυτή βρίσκεται με ένα πόδι στον κόσμο του αύριο, γιατί χρησιμοποιεί τις ικανότητάς της και έτσι μπορεί να συνδυάσει κανείς την οικογενειακή ζωή με την επαγγελματική ζωή. Έτσι λοιπόν παίρνουμε ένα πρόβλημα, το μετατρέπουμε σε σχέση με τη σύλληψή του με διαφορετικό τρόπο και περνάμε στον κόσμο της αύριο. Πολλοί δάσκαλοι λοιπόν έχουν κάνει καταπληκτικά πράγματα. Ενώ λέγαν άλλοι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει δυνατόν. Ελπίζω για τον επόμενο χρόνο που θα αρχίσει το Σεπτέμβριο του 2013 ότι θα μπορέσω να βοηθήσω αυτούς που έχουν την ανάγκη και να χρησιμοποιήσουμε τις νέες πλατφόρμες των ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για να έχουμε επικοινωνία προς όλους και να συνεχίσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες, γιατί οι πρωτοβουλίες είναι σωστές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Σάσκια. Η Μόνικ Μόροου έχει το λόγο από τη ΣΥΣΚΟ. Εγώ είμαι τεχνολόγος, είμαι γυναίκα και δεν ζητάω συγγνώμη. Εγώ βλέπετε πως κινώ το χέρι μου για να αλλάζω και εγώ τις διαφανίες μου. Αυτά που θα σας πω μέσα σε 10 λεπτά έχουν σαν νόημα τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, είτε είναι δημόσιες οι επιχειρήσεις είτε ιδιωτικές, που να είναι πρόσφορο για τις γυναίκες θα πρέπει να λειτουργήσουμε προληπτικά στον συγκεκριμένο τομέα. Είχα μία γυναίκα που με προετοίμαζε από τον χώρο τον ραδιοτηλεοπτικό και μου έλεγε ότι αν δεν γράψεις εσύ το σενάριο της σταδιοδρομίας σου και το ρόλο σου θα στο γράψουν άλλοι για σένα. Αυτό έγινε με μένα και στη ΣΥΣΚΟ τα καταφέρνουμε αλλά πάντα μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Όταν θέλουμε λοιπόν να υπάρχει ποικιλότητα στο χώρο εργασίας πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό, τι πρέπει να κάνουμε, τι στόχους πρέπει να κάνουμε. Ε, θα συνδέσουμε τα μπόνους μας σαν παράδειγμα με τους στόχους μας για την γυναίκα. Συνεπώς, το επόμενο θέμα. Έχουμε κάποιες προτεραιότητες ε, θα έλεγα επιχειρηματικές. Ε, εγώ ξέρω και το τι κάνει η Ρουθ με τη δική της επιχείρηση οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Αν δεν έχει κανείς την ποικιλότητα, ιδιαίτερα στον τομέα των φύλων, αυτό θα επηρεάσει τελικά την απόδοσή σου. Οι στατιστικές το μαρτυρούν αυτό. Θα πρέπει λοιπόν όχι να αναζητούμε τις στατιστικές, αλλά να παραδεχθούμε το ποια είναι η πραγματικότητα. Να λοιπόν κάποια πράγματα εδώ, τα οποία ξέρετε και γνωρίζετε Υπάρχει μια δυνατότητα θα έλεγα οι γυναίκες στον τομέα της τεχνολογίας να είναι πιο ορατές. Να θυμάστε όμως κάτι γυναίκες και άνδρες ότι είσαστε εσείς υπεύθυνε για τις σταδιοδρομίες σας. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε στους οργανισμούς μας είναι να δημιουργήσουμε το πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέψει να αναπτυχθούμε θα πρέπει να δούμε ποιες είναι αυτές οι κομβικές δυνατότητες τις οποίες θα επιδιώξουμε είτε μόνοι μας είτε με άλλους. Θα πρέπει εμείς να δίνουμε το παράδειγμα προς τα έξω, να θέλουμε εμείς να είμαστε πρόσωπα αναφοράς, πρότυπα αναφοράς. Αυτό θα το πετύχουμε με τον προληπτικό τρόπο. Έτσι θα γίνουμε ε, οι γυναίκες ηγέτιδες ε, στην συγκεκριμένη περίπτωση. Και έτσι θα είμαστε και πρότυπο και για τους άνδρες, όχι μόνο για τις γυναίκες. Θα πρέπει να το πετύχουμε αυτό ούσες ευαίσθητες σε σχέση με αυτά τα θέματα. Να δείχνουμε λοιπόν ποιες είναι οι γυναίκες, να είναι ορατές οι γυναίκες. Θα πρέπει επίσης ε, ε, οι συγκεκριμένες γυναίκες ε, να σχεδιάζουν οι ίδιες, αν θέλετε, τα πρότυπά τους και να αποτελούν από μόνες τους πρότυπο. Κοιτάξτε, αυτό που κάνουμε τώρα είναι ωραίο, αλλά δεν θα πρέπει να γίνεται άπαξ ή θα πρέπει να γίνεται επειδή είναι της μόδας. Εγώ συνάντησα εκπληκτικά κορίτσια σήμερα εδώ, συνάντησα πραγματικά εξαιρετικά κορίτσια και γυναίκες και έχω εντυπωσιαστεί. Λοιπόν, πού είναι οι άνδρες όμως για να τα συζητήσουμε μαζί τους. Θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία και με τους άνδρες. Θα πρέπει επίσης να είμαστε όλοι οι η Γενική Διευθύντρια της υπηρεσίας μου είναι, της εταιρείας μου είναι γυναίκα, ταυτόχρονα και η Διευθύντρια του τμήματός μου είναι γυναίκα. Πρέπει η μισή σε κάθε επιχείρηση να είναι γυναίκες. Λοιπόν, ας αναγνωρίσουμε επίσης τις γυναίκες ε, ε, την προσπάθεια την οποία κάνουν στο χώρο εργασίας τους. Δεν το έχουμε κάνει αυτό. Θα πρέπει να προωθούμε τις γυναίκες οι οποίες συνεισφέρουν στον τεχνολογικό τομέα. Εγώ έχω πολύ σημαντικές γυναίκες στην επιχείρησή μου, συναντήθηκα μαζί τους την προηγούμενη εβδομάδα, είδα τι τεράστια εξουσία. Μία έχει σπουδάσει ιατρική για κάποια χρόνια και ασχολείται με την ηλεκτρονική υγεία και πώς μπορεί να επηρεάσει ε, την υγεία των πολιτών. Οι υβριδικές ικανότητες, οι υπολογιστές και η τέχνη, οι υπολογιστές και η υγεία είναι μια τεράστια ευκαιρία. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για μας και έτσι οι γυναίκες θα φανούν περισσότερο. Αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα σε μια οργάνωση, θα πρέπει να υπάρξει σωστή κατανομή των αρμοδιοτήτων. Μία γυναίκα είπε ότι εγώ είμαι με αυτή την επιχείρηση δύο, επιχείρηση δύο χρόνια και δεν μπορώ να περιμένω πέντε χρόνια για να αλλάξω κλάδο μετά. Θέλω να κινούμε, θέλω αν ασχολούμαι με τα θέματα τροφοδοσίας ας πούμε, θα πρέπει να έχω τη δυνατότητα να ασχοληθώ με αυτά που με ενδιαφέρουν και για τα οποία είμαι εκπαιδευμένη οι γυναίκες σηκώνουν τα χέρια τους, λένε το τι θέλουν και εσείς οι γυναίκες θα πρέπει να λέτε τι θέλετε, δεν θα πρέπει να ντρέπεστε. Θέλετε θέσεις υψηλής απόδοσης, θέλετε να διευρύνετε τα δίκτυά σας. Έχουμε ήδη εξαιρετικά δίκτυα γυναικών επιχειρηματιών και άλλων στην Ευρώπη. Και από μια έκθεση McKinsey χρειαζόμαστε, δείχνει ότι χρειαζόμαστε πρότυπα και πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό όχι μόνο κάποιος ο οποίος γράφει ένα βιβλίο. Θα πρέπει να δούμε στην δουλειά με ποιους ανθρώπους μπορούμε να ταυτιστούμε. Γνώρισα μια γυναίκα από το Σαντιέγο που κάνει εξαιρετικά πράγματα σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας και της έχω ζητήσει να ενημερώσει πάρα πολύ κόσμο σε σχέση με όλα αυτά να βλέπετε επίσης και την δυνατότητα εναλλαγής θέσεων. Ξέρετε ότι είμαι πάρα πολύ σύντομη και πηγαίνω απευθεία στην ουσία. Η Grace Hopper που είναι ηρωίδα για μένα, γιατί δημιούργησε τους αλγορίθμους. Ξέρετε ότι όλοι στις δεκαετία του 40 της έλεγα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα και του 50. Παρ' όλα αυτά είχε το θάρρος να συνεχίσει, δεν δέχτηκε ποτέ το όχι και ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε λέει ότι είναι ευκολότερο να ζητά συγνώμη παρά να ζητά άδεια. Πόσες φορές έχετε πάει σε μια συνεδρίαση και λέτε κοιτάξτε θέλω να κάνω αυτό, αφήστε με να το κάνω. Όχι, να το κάνετε. Και αν μπερδευτείτε στα πόδια κάποιου άλλου γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε σε αυτή την περίπτωση ζητήστε συγνώμη αλλά είναι προτιμότερο να κάνετε αυτό που πρέπει, να παίρνετε την πρωτοβουλία και αυτό θα πρέπει να έχετε σαν στόχο. Να κάνετε αυτό το οποίο πιστεύετε εσείς ότι είναι σημαντικό. Και τέλος, πάθος. Το πάθος είναι το 50% του ε, ό,τι και να κάνουμε και να κάνετε. Ας έχετε το πάθος να προχωρήσετε λοιπόν σε αυτήν την τεχνολογία. Η θέση των γυναικών είναι πολύ σικ να προωθηθεί στην τεχνολογία που μας ενδιαφέρει. Ευχαριστούμε τις ομιλητριές μας. Τρεις παρεμβάσεις έχουν προγραμματίσει από τρεις ευρωβουλευτές που παρακολουθούν τακτικά αυτά τα θέματα. Η κυρία Χέρτζοκ είναι η πρώτη. Έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μεγάλη μέρα σήμερα για μένα. Εγώ έκανα προσπάθεια επί δύο χρόνια για να μπει αυτό το θέμα στη μέση διάταξη και χαίρομαι που έγινε πραγματικότητα. Ε, ποια ήταν η καλύτερη μου μέρα αυτή τη εβδομάδα, σε ένα λεπτό θα το πω. Τη Δευτέρα μπήκα στο Σοφιτέλ για να γνωρίσω, να συναντηθώ με τον Έτιγκερ για θέματα ε, ενέργειας. Ε, μια γυναίκα ε, με σταμάτησε και μου είπε χρησιμοποιήστε τα σλόγγαν σας. Ποιο σλόγγαν εννοείται της λέτε. Ήταν μια επιχειρηματίας που έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση ε, και την γνώρισα ε, σε μια συνάντηση που είχε γίνει με τέτοιους επιχειρηματίες. Ε, με ρώτησε τι πρέπει να κάνουμε. Της είπα ότι πρέπει να αλλάξετε το πώς μιλάτε. Αυτό το λέω και το ξαναλέω. Ε, πιστεύω ότι ο τομέας τη πληροφορική θα πρέπει να ανοίξει στι γυναίκε και να τους πει έχουμε μια προσφορά εδώ. Και ο τομέα τη πληροφορική με τι γυναίκε μέσα θα πρέπει να στραφεί προ του πολιτικού και να, πει. και να τους πει έχουμε προσφορά. Εάν θέλετε να βγείτε από την κρίση, δεν θα πρέπει να επιβάλλετε μόνο σκληρή δίαιτα, γιατί δεν χάνει κανείς βάρος με τρελή δίαιτα, αλλά πρέπει να κάνει και αθλητισμό. Η οι γυναίκες μέσα στην πληροφορική μπορεί να είναι η πλευρά του αθλητισμού για να βοηθήσει τις κοινωνίες να βγουν από την κρίση. Πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε ο τομέας της πληροφορικής με γυναίκες μέσα να ανοίξει και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, επιτρέψτε μου ακόμα μισό λεπτό να σας το εξηγήσω αυτό. Να σας πω μια ιστορία. Ένας κτηνίατρος στην ε, επικράτειά μου ε, δεν μπορούσε να στην εκλογική μου περιφέρεια δεν μπορούσε να γράψει, ε, δεν είχε καλογραφικό χαρακτήρα και άρχισε να χρησιμοποιεί το κομπιούτερ. Ε, που είναι γυναίκα. Ε, χάρη σε αυτή την... Α, χάρη αυτή την ενασχόλησή της με, την, τον υπολογιστή, έγινε γνωστή και όλοι πήγαιναν σε αυτή και έγινε ε, εκατομμυρίουχος. Ε, η εμπειρία μου με, το, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να περάσουμε από τα μικρά στα μεγάλα κατευθείαν, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεγάλες. Εδώ τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να βοηθήσουν ε, και οι γυναίκες μπορούν να βοηθήσουν πολύ, να είναι ο ενδιάμεσος κρίκος. Μπορείτε να συμφωνείτε με αυτό. Ευχαριστώ κυρία Χέρτζοκ, η κυρία Τσικάου. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα χρησιμοποιήσω τη ρουμανική γλώσσα γιατί είναι όμορφη γλώσσα και έχουμε και μετάφραση εξάλλου. Ελπίζω θα αρέσει γενικά αυτή η γλώσσα. Να ξεκινήσω συγχαίρουσα του οργανωτές ή τις οργανώτριες και κυρίως την Επίτροπο Νέλη Κρούζ εδώ και πολλά χρόνια προωθεί τη θέση των γυναικών στις τεχνολογίες ICT. Το γεγονός λοιπόν ότι είχαμε μια σειρά από εκδηλώσεις προς την κατεύθυνση αυτή καταδεικνύει ότι αρχίζουν σιγά σιγά να γυρίζουν τα γρανάζια. Θα ήθελα σήμερα να υπήρχαν και άλλα γεγονότα αυτού του είδους σε εθνικό επίπεδο. Χρειαζόμαστε πολλές γυναίκες πρωταθλήτρες της τεχνολογίας πληροφορίας σε εθνικό επίπεδο για να είναι υποδείγματα ρόλου και να βοηθήσουν τις νέες γυναίκες να διαλέξουν μια καριέρα στις επιστήμες ή στην πληροφορική. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από το δημοτικό. Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση <clears throat> για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε <clears throat> τις νέες κοπέλες να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες στα θέματα της πληροφορικής. Ξεκινώντας λοιπόν από το δημοτικό, περνώντας στο γυμνάσιο, στο πανεπιστήμιο. Χρειαζόμαστε αυτές τις δεξιότητες για να μπορέσουν οι γυναίκες αυτές να μπουν στην αγορά εργασίας. <clears throat> Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα βελτιώσουμε τα αποτελέσματα αυτά χωρίς να έχουμε πραγματική χρηματοδότηση. Νομίζω ότι μόνο με μια προορατική δράση και με την ενθάρρυνση προς τους νέους να διαλέξουν καριέρες στον τομέα της ICT που θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην ε, εξέλιξη της κοινωνίας μας. Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, θα ήθελα να ζητήσω από την Επίτροπο να συνεχίσει να αγωνίζεται για να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν καθόλου περικοπές στην διευκόλυνση Connecting Europe γιατί οποιασδήποτε τέτοιες περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στους εθνικούς προϋπολογισμούς θα σημαίνουν λιγότερη δημιουργία θέσεων απασχόληση για τους νέους και ιδίως για τις γυναίκες στις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίας. Επειδή έχουμε διάφορες ε, πολύ εξέχουσες ε, κυρίες που έρχονται από τον ιδιωτικό τομέα μαζί μας σήμερα και που ήδη <clears throat> είναι ανεγνωρισμένες στον χώρο της ICT, και στην έρευνα και στην διαχείριση επιχειρήσεων, θέλω να πω ότι θα ήταν χρήσιμο να είχαμε ένα πρόγραμμα τύπου έρασμος για τους νέους, για τις νέες κοπέλες που εργάζονται στον τομέα της ICT και προσπαθούν να δημιουργήσουν εκεί μια καριέρα. Να έχουμε υποτροφίες τύπου Εράσμου θα ήταν πολύ χρήσιμο για την επίτευξη αυτού του στόχου θα μπορούσε να γίνεται αυτό σε ευρύτερο επίπεδο από την Ευρώπη και μόνο. Έχουμε τον εκπρόσωπο της Διεθνούς Ένωσης Επικοινωνίας και εκπροσώπους παγκοσμίων εταιριών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να τονώσουμε την επαφή μεταξύ ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων και ενδιαφερομένων για τις τεχνολογίες ICT. Στη Ρουμανία υπάρχουν πολλοί νέοι οι οποίοι έχουν σπουδάσει θετικές επιστήμες Υπολογιστέ, μαθηματικά και θα ενδιαφερόντουσαν πάρα πολύ. Μιλάω για κοπέλε. Θα ενδιαφερόντουσαν πάρα πολύ να, να συμμετάσχουν σε τέτοιε πρωτοβουλίε. Οργανώσαμε μια τέτοια διάσκεψη για την πληροφορική στη Ρουμανία και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τούρα για το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό να πείσουμε τις γυναίκες ότι μπορούν να γίνουν πράγματα στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Il... Ακούσουμε έναν άνδρα τώρα, τον κύριο Κέλλη. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τις ομιλήτριες. Όταν ήρθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και τέσσερα χρόνια, μου έκανε εντύπωση ο μεγάλος αριθμός των γυναικών ήταν πολύ περισσότερο από αυτά που είχα δει στη χώρα μου, είτε στην Βουλή της Ιρλανδίας, είτε στους Δήμους κτλ. Είμαι σε τρεις κοινοβουλευτικές επιτροπές και στις τρεις προεδρεύουν γυναίκες. Εδώ είστε εσείς πρόεδρος, η τα Χούντμπερ, επίσης την άλλη και η Ντόρις Πακ στην εκπαίδευση, πολιτισμό και αθλητισμό. Αναφερθήκατε επίσης ε, κυρία Μόρου ότι καλύτερα να ζητά συγγνώμη κανείς παρά άδεια. Ε, η κυρία Πακ που είναι πρόεδρο στην Επιτροπή Πολιτισμού ούτε το να κάνει ούτε τα άλλο και όμως τα πράγματα γίνονται όπως αυτή θέλει. Είναι και αυτός ένας τρόπος και πολλοί από τους επιτρόπους επίσης είναι ε, γυναίκες, εξαιρετικοί επίτροποι όπως η κυρία Κρούς, η Ιρλανδή επίτροπος, η κυρία Κουίν γενικά. Νομίζω ότι δέχονται τις γυναίκες και προωθούν τις γυναίκες και δεν χρειάζεται να τους καταλογίζουμε αρνητικά. Τώρα σχετικά με το Connecting Europe θα ήθελα να δούμε τι γίνεται σε σχέση με, την, ε, με το ευρύ φάσμα γιατί από ό,τι φαίνεται ο προϋπολογισμός θα μειωθεί μέχρι και 90%. Ελπίζω να μην γίνει. Αν τυχόν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι καταστροφικό για αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Επίτροπε, αναφερθήκατε κι εσείς και στη συγκεκριμένη επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε στο Κόρκ από τον Μπάντον και τον Λίο μια υπηρεσία η οποία καθοδηγεί τα νέα παιδιά από 6 ετών μέχρι 16 ετών έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν συγκεκριμένες ικανότητες. Ελπίζουμε 2 εκατομμύρια θέσεων που δεν μπορούν να πληρωθούν στην Ευρώπη λόγω έλλειψης ε, ικανοτήτων, αυτό να το αλλάξουμε και να το διορθώσουμε. Ξεπέρασα το χρόνο μου, δεν θα πρέπει να, αφήσω άλλες γυναίκες να μιλήσουν. Riera Madurell, prego. Muchas gracias, Presidenta. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες για τον ενθουσιασμό που έχουν δείξει, για τις εξηγήσει. Και εμείς αγωνόμαστε πάντα γι' αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε γυναίκες με τόσο ενθουσιασμό και τόση δυναμικότητα. Και πριν από όλα αυτά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις διοργανώτριες αυτής της εκδήλωσης, και ιδιαίτερα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και στην Επίτροπο. Και ξέρω ότι η Επιτροπή Ήτρα έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μας ενδιαφέρει και το θέμα της έρευνας και της ε, καινοτομίας. Και ίσως για πρώτη φορά η πρόταση της Κομισιόν για ένα νέο πρόγραμμα στο πρόγραμμα πλαίσιο Ευρώπη 2020 υπάρχει και ένα τμήμα που έχει να κάνει με τη διάσταση του φύλου που το Κοινοβούλιο το έχει ταλαιπωρήσει λιγάκι, ε, είχε να κάνει με ένα σωστό ποσοστό για τη συμμετοχή των γυναικών. Αυτό ήταν πολύ θετικό. Νομίζω ότι αυτό είναι χρήσιμο να υπάρχει και να τονίσουμε ότι υπάρχει στο πρόγραμμα πλαίσιο. Θέλω λοιπόν να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία να εκφράσω δημόσια την ευγνωμοσύνη μου. Επίση όμω θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα. Άκουσα πολλά πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα μπορούν να ισχύουν για πολλού τομεί και ιδίως στις επιστήμες, στην έρευνα. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα τομέα που έχει κάποιες ιδιοτυπίες. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι στα σχολεία, τα καλά σχολεία γενικά, υπάρχουν πάντα τα θέματα αυτά των τεχνολογιών της ε, πληροφορίας και των επικοινωνιών, αλλά όλα αυτά είναι τα ίδια για τα αγόρια και τα κορίτσια. Υπάρχει αρκετή ισότης καταρχήν. Αυτό το οποίο εμένα μου κάνει εντύπωση ότι τα 90% των κοριτσιών ενδιαφέρονται για τα ε, επιστημονικά θέματα. Φαίνεται λοιπόν ότι η ρήξη, η τομή γίνεται κάπως αργότερα. Βλέπουμε στα πανεπιστήμια ότι φυσικά είναι πολύ μειωμένο το, το ποσοστό των γυναικών και στο χώρο εργασίας. Ξέρουμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία που μας αναφέρατε και φυσικά οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται πάρα πολύ να υπάρχουν και οι γυναίκες στο χώρο εργασίας και της ε, επιστήμης. Δεν θέλουμε να σπαταλάμε τους μισούς εγκεφάλους στην κοινωνία μας. Είναι λοιπόν και οικονομικό το συμφέρον για αυτές τις ενέργειες. Εμείς λοιπόν Θέλουμε να μελετήσουμε καλύτερα τις αιτίε για αυτήν τη διαφορά που παρατηρείται μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Και νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι η Κομισιόν μπορεί αυτό να το ενσωματώσει στις νέες έρευνες που θα κάνει. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω λίγο καλύτερα πού βρίσκονται οι ιδιαιτερότητες αυτού του τομέα των ε, τεχνολογιών ICT. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που σας περιορίζω. αλλά κάθε φορά ξεχνάω να ελέγχω τα προγράμματα και τελικά πάντα βάζουμε πολλούς ομιλητές και με αναγκάζουν τελικά όταν έρχεται η ώρα να σας πιέζω ε, με τρόπο απαράδεκτο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα δώσω ένα-δύο λεφτά στον καθένα, όχι παραπάνω, γιατί δεν έχουμε παραπάνω, στους ε, ομιλητές μας για να απαντήσουν στις ερωτήσεις ε, και τις παρατηρήσεις που άκουσα. Ποιος θέλει να ε, ξεκινήσει η Τζάνα Μαρτινέγκο. Ναι, να δώσω κάποιες απαντήσεις. Καταρχάς, ο κατακαιρματισμός των επιχειρήσεων πληροφορικής, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το, στην Ιταλία το 90% των επιχειρήσεων πληροφορικής έχουν τέσσερις υπαλλήλους. Αυτό καθιστά την πορεία τους πολύ περίπλοκη και πρέπει να ξαναδούμε εντελώς ε, τη σχέση μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων. Αυτό το σενάριο που ακούστηκε, να δημιουργήσουμε μια κινητικότητα μεταξύ των νέων, μιλάω για τη Ρουμανία, έτσι, και τις επιχειρήσεις, με μια ανταλλαγή, ας πούμε, και μια ε, συνοδεία, παύλα μαθητεία, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Είναι μια εμπειρία που έζησα και εγώ έμεσα ε, στην Ακαδημία Βουλιαρική Ακαδημία Επιστημών και στην ε, Ρουμανία επίση το ζήσα. Είναι χώρες και υπάρχουν και πολλές τέτοιες χώρες στην Ευρώπη μας που θεωρούνται από τι επιχειρήσεις όπου ε, είναι ελκυστικέ χώρες για να μετεκατασταθούν οι επιχειρήσει τους. Έτσι τις βλέπουν οι επιχειρήσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να ανακτήσουμε αυτό το ανθρώπινο δυναμικό με την κινητικότητα και με την πλαισίωση και την ε, βοήθεια που θα δώσουμε σε αυτούς του ανθρώπους καθ' όλη τη διάρκεια τη πορεία. του Ευχαριστώ. Η κυρία Σάσκια. Δύο λεπτά, τρία σημεία. Εγώ είμαι πρόεδρος του Συμβουλίου μιας επιχείρησης της πληροφορικής. Το 50% αυτών που δουλεύουν στην Πουλ δεν έχουν κάνει σπουδές τεχνολογίας. Έχουμε ακόμα και γυμναστές αλλά έτσι και αλλιώς ε, ο αθλητισμός βοηθάει στην υγεία των εργαζόμενων στον τομέα. Λοιπόν, έχουμε προβλήματα μόνο σε ακραίες καταστάσεις. Στην επαγγελματική μου ζωή, ε, στην ε, Μπουλ, έχουμε ακόμα και αναλυτές σε σχέση με ακραία σενάρια αν είναι πραγματιστής, αν κάποιος έχει ασχοληθεί ας πούμε με εγκληματολογία και πρέπει να κάνει μια τέτοια ανάλυση στον τομέα της αστυνομίας, τότε προφανώς και έχει τα προσόντα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι πρέπει να έχει τεχνολογικές ικανότητες, πρέπει να έχει ηγετική στάση, πρέπει να έχει πάρα πολύ καλές αναλυτικές ικανότητες και φυσικά οι γυναίκες είναι σε θέση να κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί πολλές φορές δεν θα πετύχουμε τις επιθυμητές λύσεις. Να κινητοποιήσουμε λοιπόν την ανάπτυξη, αλλά να προχωρήσουμε και με έξυπνες ευφυείς μελέτες και εφάνταστες και καινοτόμες προσπάθειες. Και έτσι θα δώσουμε κίνητρα στις γυναίκες, ανεξαρτήτως των σπουδών τους, να προχωρήσουν. Οι γυναίκες σπουδάζουν όχι για να έχουν μια επαγγελματική ζωή, αλλά σπουδάζουν γιατί θέλουν να αποκτήσουν κάποια ειδικά χαρακτηριστικά. Στο Βέλγιο, σαν παράδειγμα, το να μην κάνεις τίποτα μετά από το μάστερ ή να κάνεις ένα μάστερ μετά το μάστερ είναι πάρα πολύ ε, συνηθισμένο. Κάνουν ένα μάστερ ιστορία γιατί τους ενδιέφερε και μετά κάνουν ένα μάστερ γλώσσας. Λοιπόν, έτσι ε, εκμεταλλεύεται κανείς τα πανεπιστήμια. Δεύτερον, 15 εβδομάδες στάζ, όπως λένε στα γαλλικά, στην επιχείρησή μου τότε εγώ θα ενδιαφερόμουν για κάτι τέτοιο. Είναι ιδανικός τρόπος για να πιστούν οι γυναίκες αυτές που έχουν κάνει σπουδές ότι ο πραγματικός κόσμος είναι διαφορετικός αλλά είναι cool και αστείος. Αν μου φέρεις κάποιον για τρεις μέρες τότε εγώ το μήνυμα αυτό δεν μπορώ να το περάσω. Δεν μπορώ να εμφυσίσω τον ενθουσιασμό. Νομίζω ότι είναι βάρος για την εταιρεία και είναι και μειονέκτημα για το συγκεκριμένο πρόσωπο. 15 εβδομάδες λοιπόν τα στάζουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουν και οι φοιτητές, οι σπουδαστές να γνωρίσουν ποια είναι η πραγματικότητα. Τώρα για τις γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει κάποιες ε, σπουδές τεχνικές αλλά δεν ασχολούνται με τον τομέα τους μετά. Έθεσα το θέμα με διαφορετικό τρόπο στις γυναίκες της Μπουλ. Μου είπαν γιατί ήρθατε εδώ. Μου απάντησαν ότι ήρθαμε εδώ γιατί είχαμε κάποια χρόνια στην ουσία δυνατότητα σε σε ένα κλαμπ ανδρών, σε ένα κλαμπ αγοριών. Και μετά έπρεπε να επιμείνουμε, να φανούμε ζόρικες, γιατί όπως είπα στην αρχή, δεν ήξερα ακριβώς πώς θα μπορούσα να συνεισφέρω στο να δοθούν απαντήσεις στα ερωτηματικά για τη ζωή. Και τώρα μετά από κάποια χρόνια άρχισα να κατανοώ ότι το δικό μου κομμάτι αν το βάλω στο πάζολ στη σωστή θέση τότε θα βρεθώ στο κέντρο της λύσης. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Η προσωπική εμπειρία έχει σημασία, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι που σπουδάζουν, οι γυναίκες που σπουδάζουν, ναι μεν σπουδάζουν αλλά δεν ξέρουν για πού θα πρέπει να κατευθυνθούν μετά. Ευχαριστώ πραγματικά. Σας δώσαμε, ε, μας λιτώσατε και μισό λεπτό γιατί μίλησατε μόνο ένα μισό λεπτό. Κυρία Μόρου, σύντομα. Ε, κάτι προσωπικό. Η κυρία Κρούς το ξέρει. Ε, η προσωπική μου ιστορία αφορά το θάρρος. Όταν έφτασα πρώτη φορά στην ε, Ελβετία, μου έδωσε, το αφεντικό μου έδωσε ένα βιβλίο για το Μακιαβέλη. Και ουσιαστικά έμαθα ότι αν θες να προχωρήσεις σε μια οργάνωση θα πρέπει να μάθεις κάποια πράγματα. Καταρχάς θα, θα έπρεπε να είσαι συντηρητικός, θα έπρεπε να είσαι παντρεμένο, δύο παιδιά, δυόμιση μάλλον παιδιά. Το μισό ήταν ε, εικόσιτο. Θα πρέπει να τα πας καλά και να ανήκει στον Ελβετικό στρατό. Ήταν η πρώτη μου δουλειά, η πρώτη μου μέρα στη δουλειά, έτσι. Και τότε τα μάθα αυτά και έμαθα πάνω απ' όλα ότι δεν πρέπει να είσαι γυναίκα. Αλλά όλα αυτά με έκαναν να συνεχίσω. Ε, μπορούμε να σας δώσουμε πολλές ε, συνταγές ε, για το πώς θα επιτύχεις. Αλλά πώς θα τα καταφέρεις. Εδώ βρίσκεται η επιτυχία, στην κοιλιά σου μέσα, στα εντόστια σου. Ε, μπορείς να πας σε διάφορες σχολές, σε διάφορα πανεπιστήμια έτσι, τεχνολογικά κτλ. Και βλέπεις μέσα στις τάξεις δύο κορίτσια. Ε, εγώ θα... Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τομέας, συμφωνώ με τη Σάσκια. Ε, γιατί και εγώ ε, ξεκίνησα από τελείως αλλού. Ξεκίνησα από την γαλλική φιλολογία. Δεν σπούδασα μηχανική, μηχανικός, έτσι. Το, βασικό είναι να έχει κανείς α, τη σωστή αντίληψη στον 21ο αιώνα. Ευχαριστώ πραγματικά. Και τώρα η Επίτροπος έχει τον λόγο. Θε, πρόεδρε σκέφτομαι ένα γεγονός. Όλοι μας έχουμε Οι γυναίκες μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 89 με τις τελευταίες στατιστικές. Και γι' αυτό εγώ ίσως είμαι υπερβολική στη χρήση αυτού του ε, Παραδείγματο ακόμα και αν σας εντυπωσιάζει ένας πρίγκιπας ο οποίο έρχεται με το άσπρο του άλογο μπορεί να εξαφανιστεί μετά. Εγώ πάντως έχω μια εμπειρία. Πρέπει να ζει κανείς με ένα πρίγκιπα ή έστω με ένα φίλο, ένα σύντροφο για άλλο λόγο από το να τον αγαπάει κανείς και να εξαρτάται από αυτόν. Όχι, πρέπει να πάρετε τη δικιά σας γραμμή στη ζωή. Και οι εγκέφαλοι των γυναικών μπορεί να φταίνε. Δεν μπορείτε να τα έχετε όλα στη ζωή. Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι αν έχετε αυτόν τον σύντροφο, είτε ένα άνδρας ή γυναίκα ή οτιδήποτε, αν θέλετε να έχετε μια οικογένεια, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η οικογενειακή ζωή δεν είναι παρά μόνο ένα μικρό κομμάτι της ζωής. Θα πρέπει να έχετε την δική σας ζωή. Σάσκια, εσύ είσαι πολύ ανοιχτή σε αυτά τα θέματα. Έχεις πέντε παιδιά, έχεις μια καριέρα Τέσσερα. Τέσσερα πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Και ξέρω ότι πρέπει να πάρει δύσκολε αποφάσει πολλέ φορέ. Όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται σε αυτές τις καταστάσεις. Υπάρχουν στιγμέ. που έχω πέρασει και εγώ τέτοιε δυσκολίε και νομίζω ότι πήρε τη σωστή θέση, έκανε τις σωστές αντιδράσεις σε αυτές τις στιγμές. Αλλά όταν μιλάμε για υποδείγματα ρόλου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περιπτώσει όπως η Σάσκερ. Δεν είναι η καριέρα ή η οικογένεια, όχι. Μπορείτε να τα καταφέρετε και τα δύο, αλλά χρειάζεται θάρρος και στένος. Τούτου λεχθέντος. σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν οι γυναίκες. Πριν και μετά τα παιδιά πρέπει να δίνουμε έμφαση στην ε, σταδιοδρομία σας. Δεν θα πρέπει να την παραμελείτε την ε, σταδιοδρομία σας. Πρέπει να παίξετε ηγετικό ρόλο και σε αυτό το τομέα και όχι μόνο στην οικογένεια. Είναι μια κατάσταση όμως που σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερα υποδείγματα ρόλου από τις γυναίκες που αριστεύουν στον τομέα τους, όσο περισσότερα αυτά τα μοντέλα ρόλου, τόσο πιο πολύ θα πρέπει να τις, να τις εξάρουμε και να τις προβάλλουμε. Για δύο ερωτήσεις που τέθηκαν από τα μέλη του Κοινοβουλίου. Δείχνουν όλα αυτά ότι είμαστε παρασάγκας από το τι λέει η κυρία Κρούζ. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες για το Connecting Europe, αλλά ένα πολύ μικρό τμήμα αυτού του Horizon 2020, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένα πρόγραμμα επταετούς χαρακτήρα που ξεκινά από το επόμενο έτος. Μα ακόμα και οι κομμουνιστές δεν κάνανε ετή προγράμματα ετή ήταν το μάξιμο που καταφέρανε. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πενταετή προγράμματα. Εν πάση ένα τμήμα του προπολογισμού αυτού έχει προσδιοριστεί για επενδύσεις που δεν είναι ελκυστικά για τον ιδιωτικό τομέα. Και επομένως το παράδειγμα αυτό το οποίο ανέφερε η Σάσκια δεν θα πρέπει να χωρίσουμε την κοινωνία μας σε δύο τμήματα, αυτούς που έχουν και αυτούς που δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι δεδομένο αυτό, ότι κάποιοι θα έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες και κάποιοι όχι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο σφάλμα, δεν πρέπει να το αποδεχτούμε. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε με την <clears throat> Connecting Europe Facility. Μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα κτλ. αλλά οι ηγέτες των 27-28 σύντομα κρατών μελών πήραν μια απόφαση ότι δεν πρέπει να φυγούν αυτά τα κονδύλια, τα 9 δισεκατομμύρια. στους τομείς αυτούς όπου ότι δεν μπορούν να δαπανηθούν μάλλον τα χρήματα που χρειάζονται για να αντισταθμίσουν της, την έλλειψη ιδιωτικών πρωτοβουλειών. Η μόνη μου ελπίδα είναι ότι το Κοινοβούλιο με την σοφία του θα ανατρέψει την απόφαση του Συμβουλίου. Γιατί εδώ μιλάμε για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και αν δεν μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι στη μελλοντική οικονομία της Ευρώπης θα υπάρχει υποστήριξη όλων και όχι για τους λίγους, τότε κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Και επομένως όλα αυτά στα χέρια του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ Επίτροπε. Όλες γνωρίζουμε ότι έχουμε συναδέλφους που εμπλέκονται σε αυτά τα θέματα άμεσα και προσπαθούμε να επηρεάσουμε και τον προϋπολογισμό για προς την κατεύθυνση αυτή. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα πετύχουμε. Να περάσουμε τώρα στη δεύτερη σειρά, αν θέλετε, τη συνάντηση, στο δεύτερο γύρο Κίκη Στρίντ, Φάμερ, Μέτσλαρ και Τάμπορ. Ecco, voi Γνωρίζετε ότι στις 5 που θα είναι 7 στο Σαν Φρανσίσκο, θα υπάρξει ο χαιρετισμό από πλευράς της κυρία Σάντμπεργκ, η οποία είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Facebook. Λοιπόν, ξεκινάμε για να προλάβουμε λίγο την καθυστέρηση. Δίνω το λόγο στην κυρία Κίκη Στρίδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ε, Γυναικών στις Επιστήμες και την Τεχνολογία. Ευχαριστώ. Καταρχάς σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. πρώτη φορά έρχομαι εδώ και απευθύνω το λόγο. Εκπροσωπώ αν θέλετε τις γυναίκες που δουλεύουν στη βάση ε, οι γυναίκες στις επιχειρήσεις, οι γυναίκες ε, στην καινοτομία σαν εκπρόσωπος της WITEC. Τα πράγματα λοιπόν λειτουργούν με μαζικό τρόπο. Εδώ με το που σηκώνω το δάχτυλο αλλάζουν. Να μιλήσω λίγο για την οργάνωση την οποία εκπροσωπώ σήμερα, τη WITEC. Θα ήθελα να επανέλθω στα βασικά δηλαδή να σας μιλήσω για τη σημασία που έχει η υποστήριξη των γυναικών στον χώρο που μας ενδιαφέρει. Ελπίζω έγκαιρα να τελειώσω με κάποια συμπεράσματα. λοιπόν είναι ένα δίκτυο. Οι γυναίκες ε, στην επιστήμη, τη μηχανική και την τεχνολογία. Ξεκινήσαμε με την Αγγλία πολύ νωρίτερα. Σε εννέα χώρες έχουμε εκπροσώπους εταίρους και αυξάνεται ο αριθμός αυτός. Όλο και περισσότερες χώρες ετοιμάζονται να μπουν. Εργαζόμαστε σε πάρα πολλά επίπεδα για να προωθήσουμε τις σταδιοδρομίες των γυναικών στον τομέα της μηχανικής και της τεχνολογίας. Έχουμε κάνει αρκετές προσπάθειες, υπάρχουν πολλά προγράμματα μέχρι σήμερα και τη στιγμή που εμείς είμαστε εδώ διεξάγεται μία δραστηριότητα στη Σουηδία. Υπάρχει ένα workshop το οποίο συγκεντρώνει την προσοχή τους στις γυναίκες άνω των 50 ετών, οι οποίες δεν είναι πάρα πολύ ενήμερες για τα πρακτικά της τεχνολογίας των υπολογιστών, της πληροφορικής τα νέα παιδιά και οι νέοι γενικότερα είναι πολύ πιο ενήμεροι σε σχέση με την χρήση των μέσων της πληροφορικής της τεχνολογίας. Χρηματοδοτείται από την Κρούτβικ και τα κορίτσια, οι γυναίκες μαθαίνουν να διδάσκουν σε μεγάλες γυναίκες να χρησιμοποιούν πρακτικά τους υπολογιστές όπως υπηρεσίες στον τομέα των τραπεζών, αγορές α, ηλεκτρονικές και τα λοιπά, χρήση του Skype, είναι κάτι το πάρα πολύ πρακτικό και χρήσιμο. Υπάρχουν πρακτικά παραδείγματα, υπάρχουν και θεωρητικά βέβαια. Ε, πολλά είναι τα μαθήματα που δίδουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει να πω επίσης ότι η WITEC εδώ και πολλά χρόνια δραστηριοποιείται σε αυτό το κλάδο και γι' αυτό έχουμε συλλέξει θα έλεγα εξαιρετικές εμπειρίες και νομίζω ότι μπορούμε να αποτελούμε ένα πολύ σημαντικό μέσο για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορικής. Στην ουσία τώρα θα περάσω σε μία σύντομη αλλά και απογοητευτική θα έλεγα παρουσίαση του πεδίου της πληροφορικής τεχνολογίας στην Σουηδία. Διαπιστώνει κανείς, σύμφωνα με αυτό που δείχνουν οι στατιστικές, εφόσον χρησιμοποιήσουμε τις στατιστικές για να εξηγήσουμε το κατεπήγον του προβλήματος που έχουμε. Γιατί όπως είπα και όπως φαίνεται και σε αυτή τη διαφάνεια, όταν βλέπει τον τομέα στη Σουηδία, διαφέρει από άλλους τομείς. Είναι σαφές ότι υπάρχει πραγματικά ένα μεγάλο κενό, μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες. Υπάρχει ένας διαχωρισμός και διακρίσεις οριζόντια, υπάρχουν πολύ λιγότερες γυναίκες, υπάρχει κάθετη διάκριση και διαχωρισμός. Ε, οι γυναίκες όταν έρχονται να δουλέψουν σε επιχειρήσεις δεν φτάνουν σε υψηλά επίπεδα και υπάρχει και εσωτερική διάκριση όπου άνδρες και γυναίκες που έχουν τις ίδιες ικανότητες επαγγελματικές κάνουν διαφορετικά πράγματα και ακολουθούν διαφορετικούς προσανατολισμούς. Έχω εδώ επίσης όπως σας είπα κάποιες στατιστικές γιατί από τη μία έχουμε τα ψέματα και από την άλλη τις στατιστικές όπως είπε και η προλαλήσασα. Πάντως καλό θα είναι μέσα από τις στατιστικές να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς οι αριθμοί αυτοί καθορίζουν και επηρεάζουν το μέλλον μας. Νομίζω ότι η εικόνα αυτή λέει πολλά. Βλέπουμε εδώ μια δεκαετία, κάτι πάνω από μια δεκαετία ε, φοιτητών που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο στα προγράμματα ακριβώς της ε, τεχνολογίας της πληροφορικής. Όταν βλέπετε τι γινόταν το 1998 υπήρχαν λιγότερες ε, γυναίκες από άνδρες. Αλλά τι έχει συμβεί από τότε. Οι γυναίκες παραμένουν πάντα σε χαμηλό επίπεδο. Ο αριθμός των ανδρών έχει αυξηθεί τα προγράμματα έχουν αυξηθεί επίσης και βλέπετε ότι το κενό ανάμεσα στους δύο αυξάνεται. Ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε άλλου τύπου σπουδές ακαδημαϊκές. Αυτό είναι ένα ειδικό χαρακτηριστικό του τομέα της πληροφορικής, αφορά τις γυναίκες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούμε. Τι σημαίνει αυτή η διαφορά ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες θα έχει, τι ρόλο θα παίξει στο μέλλον αυτή η διαφορά. Ένα άλλο σημείο ενδιαφέρουσων στατιστικών που προέρχονται από τις επίσημες σουηδικές στατιστικές μπορούμε να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Βλέπετε τις στατιστικές για τα αποτελέσματα των εξετάσεων στον τομέα ε, της πληροφορικής για τους πολιτικούς μηχανικούς. Βλέπετε ότι εδώ και 10 χρόνια οι γυναίκες είχαν ένα μεγαλύτερο ποσοστό θετικής ανταπόκρισης στις συγκεκριμένες εξετάσεις από ό,τι σήμερα. Πολύ πιο σημαντικό από ό,τι σήμερα. Αυτά μας δείχνουν οι αριθμοί λοιπόν οι γυναίκες αναλαμβάνουν λιγότερο σημαντικές δουλειές. Και αυτό είναι αντίθετο με άλλες τάσεις στον τομέα των πανεπιστημιακό. Γιατί ειδικά στους υπολογιστές τα πράγματα είναι τόσο άσχημα για τις γυναίκες. Όποιος δουλεύει σε αυτό το χώρο, στον πανεπιστημιακό, ακαδημαϊκό χώρο, αντιμετωπίζει πάρα πολλά εμπόδια οι γυναίκες που δουλεύουν. Αν βλέπει κανείς ε, τους ανθρώπους οι οποίοι εξετάζονται στις αριστερές στήλε και τους ρωτήσετε μετά από πάρα πολλά χρόνια έχετε γίνει καθηγητές, και αυτό έχει σημασία εδώ γιατί βλέπετε ότι για τις γυναίκες είναι πολύ δύσκολο να έχουν ικανοποιητικές θέσεις ε, στις ακαδημαϊκές σπουδές. οι θέσεις για τις γυναίκες δεν είναι καθόλου μα καθόλου άνετες. Τα πανεπιστήμια δεν είναι χώροι οι οποίοι να είναι πολύ δεκτικοί για τις γυναίκες στη Σουηδία. Άλλη μία στατιστική πληροφορία για τη διάρκεια της ε, ζωής στην εργασία. Και εδώ ήρθα σε επαφή με ειδικού στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορικής. Προσπαθούμε να δούμε πόσοι εργάζονται σε τέτοιες ε, σε παροχής υπηρεσιών. Κοιτάξτε τα ποσοστά των γυναικών, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ χαμηλά βάζω και τα αποτελέσματα για την περιφέρεια της Στοκχόλμης και για το σύνολο της χώρας. Βλέπετε ότι έτσι και αλλιώς οι γυναίκες είναι λίγες, λιγότερες και δεν είναι και ιδιαίτερα εξειδικευμένες. Και όσο ψηλότερες είναι οι θέσεις τόσο λιγότερες είναι οι γυναίκε. Αυτό είναι ένα σοβαρό μειονέκτημα. Αν θέλετε όμως το πιο ανησυχητικό ε, δείχνεται από τον συγκεκριμένο αυτό ε, πίνακα. Λυπάμαι που δείχνω τόσα πολλά στατιστικά γιατί τα στατιστικά ομιλούν τη δική τους γλώσσα που είναι κατανοητή και μας λέει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Αν δείτε λοιπόν την κατάσταση για τις γυναίκες σήμερα και δείτε για τους ειδικούς τι γίνεται στους υπολογιστές, βλέπετε τις ηλικίε. Η τελευταία στήλη δείχνει το ποσοστό των γυναικών. Και βλέπετε ε, στις διάφορες ηλικιακέ περιόδους ε, τα ενδιαφέροντα των γυναικών. Οι νέες γυναίκες δεν ενδιαφέρονται, τα κορίτσια δεν ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον τομέα μας. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. οι νέες γυναίκες δεν συμμετέχουν εν πολύ στις προσπάθειες αυτές. Δεν νιώθουν άνετα στους χώρους αυτούς. Δεν ελκύονται ε, οι γυναίκες στους χώρους αυτούς. Όχι ότι δεν έχουν τις δυνατότητες, αλλά οι χώροι δεν τους προσελκύουν. Δεν τις προσελκύουν. Λοιπόν, συμπερασματικά οι γυναίκες δεν κυριαρχούν, οι άνδρες κυριαρχούν στο χώρο αυτό. Οι νέες γυναίκες δεν ακολουθούν προγράμματα στο Λύκειο και στο Πανεπιστήμιο για τους υπολογιστές. Δεν συμμετέχουν σε εξετάσεις για αποκτήσεις πιστοποιητικών ικανότητας. Και οι στατιστικές δείχνουν ότι ακόμα και αν δραστηριοποιηθούν στο συγκεκριμένο χώρο πληρώνονται λιγότερο από τις γυναίκες. Αυτά. Ήταν μια σύντομη εικόνα, πήρατε κάποια στοιχεία, μπορείτε να τα σκεφτείτε. Η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική για την παρουσία των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορικής. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. ο λόγος την Διευθύντρια Στρατηγικών Πρωτοβουλειών στο Εθνικό Κέντρο για τις Γυναίκες και την Πληροφορική. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που με προσκαλέσατε. Ακούσαμε τις στατιστικές και ε, εγώ έχω να σας προτείνω μία λύση σε αυτό το πρόβλημα. Είναι ανησυχητικές στατιστικές, έχω να πω ένα τμήμα της λύσης. Ε, Στι ΗΠΑ η κατάσταση είναι αντίστοιχη. Έχουμε πρόβλημα με τι γυναίκε και την τεχνολογία και τα κορίτσια. Το 19% των ανθρώπων που ε, είναι γυναίκες στις τεχνολογίες ε, και 18% τεχνολογικά πτυχία πηγαίνουν στις γυναίκες ε, έχει μειωθεί το ποσοστό σχέση με παλιότερα ε, και οι γυναίκες οι οποίες δουλεύουν στους τεχνικούς κλάδους παρατάνε τη δουλειά τους ε, σε διπλάσιο ποσοστό από ότι οι άντρες στο διπλάσιο της, ε, στο μισά της καριέρας τους. Ε, η απομόνωση είναι μεγάλος λόγος. Ε, αισθάνονται μόνες τους ε, οι γυναίκες στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο. τα περισσότερα σχολεία δεν, κάνουν, δεν είναι τέτοια μαθήματα και μέχρι να φτάσουν στο πανεπιστήμιο δεν ξέρουν ότι υπάρχουν τέτοια μαθήματα. Επίση δεν έχουν και πρότυπα γυναικεία. Μόνο το 11% των μηχανικών ε, ή τα ύψιλον είναι γυναίκε, επομένω δεν έχουν τα πρότυπα. Συχνά τα πρότυπα των γυναικών στην πληροφορική, όπως περνάνε από τα μέσα, είναι στερεότυπα και περνάνε το λάθος μήνυμα. Επομένως, ε, οι γυναίκες παρουσιάζονται ως καταναλωτέ τη τεχνολογία και όχι δημιουργοί της τεχνολογίας. Υπάρχουν στερεότυπα για τη γυναίκα που είναι απλώ ε, βοηθό των φυτών που φτιάχνουν τεχνολογία, και όταν δεν την παρουσιάζουν με άλλα στερεότυπα, την παρουσιάζουν ε, σαν ε, καταναλώτρια απλώς τεχνολογίας. Ε, και ούτως ή άλλως, ακόμα και αν γκουγκλάρεις τη λέξη κορίτσι, ας πούμε, μπορεί να βγάλει πορνογραφική εικόνα το ίντερνετ. Ε, ένας καθηγητής μου είπε ότι ε, ένας φοιτητής ε, φορούσε ένα μπλουζάκι της IBM ήταν μαζί με το φίλο της, ε, φορούσε ε, αυτό το μπλουζάκι που έλεγε IBM και, ποιος, και της είπε ένας καθηγητής ποιος ασχολείται με τεχνολογία, εσύ ή ο φίλος σου. Λέει εγώ, εγώ φοράω το μπλουζάκι. Α, νόμιζα ότι φοράς το μπλουζάκι του φίλου σου, της λέει αυτός. Λοιπόν, Έχω μια αντίστοιχη προσέγγιση με αυτά που ακούσαμε πριν και εμείς στον NCWTIC ε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αφύπνιση, να βρούμε τα εργαλεία κτλ. Ε, είμαστε οργανώσεις δικτυωμένες ε, στα πανεπιστήμια, στις εταιρείε, οργανώσεις εργοδοτών και ομάδες γυναικών που ασχολούνται με τεχνολογία. 450 ε, ε, οργανώσει τέτοιες έχουμε στι ΗΠΑ. Όταν εγώ μπήκα ε, σε αυτήν την οργάνωση το 2008, είμαστε πολύ λιγότεροι, αναπτυσσόμεθα και το υλικό μας αλλάζει συνέχεια. Δημιουργούμε πόρους, εν συνεχεία τους δίνουμε, τους διαδίδουμε. Ε, όλο το υλικό μου ε, είναι δωρεάν και υπάρχει online και τίποτα το θέλει μπορεί να το κατεβάσει. Ε, έχουμε πολλά προγράμματα από την αρχή ως το τέλος, από το λίκνο στον τάφο όπως λέμε. Ε, δύο από τα κορίτσια που βλέπετε στη φωτογραφία είναι και εδώ. Ε, προσπαθούμε να μιλήσουμε για τις φιλοδοξίες στον κλάδο, ε, να μιλήσουμε στις γυναίκες. Χρησιμοποιούμε αυτές τις 405 οργανώσεις του δικτύου για να εντοπίσουμε, να αναγνωρίσουμε και να υποστηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε τις νέες γυναίκες στη τεχνολογία. Ε, η πρώτη φάση είναι να βρούμε αυτές τις γυναίκες. Σε συνεχεία τα κορίτσια μας που βρίσκονται στο, στο γυμνάσιο αυτή τη στιγμή ενδιαφέρονται για τεχνολογία, αλλά 60% από αυτές θα διαλέξουν διαφορετική η κατεύθυνση στο πανεπιστήμιο. Ε, δηλαδή, ακόμα και τα κορίτσια που τα έχουμε, που τα έχουμε κερδίσει στην ε, οργάνωσή μου, δεν θα τα κρατήσουμε. Το, επομένως, η θεωρία μου για την αλλαγή είναι να κρατήσουμε αυτές τις ε, κοπέλες και, και να τις χρησιμοποιήσουμε ως μοχλό για να πείσουμε και τις υπόλοιπες κοπέλες. Ε, γι' αυτό τι κάνουμε, χρησιμοποιούμε ένα βραβείο. Ε, ε, το βραβείο το πήρε μια κοπέλα και λέει ε, αυτό το βραβείο δείχνει ότι αρκετά, έχω αρκετή εμπιστοσύνη στον εαυτό μου για να διαλέξω μια τέτοια κατεύθυνση στο πανεπιστήμιο. Εδώ βλέπουμε ε, γυναίκες ε, που έχουν διευθυντικέ θέσει στη Μοτορόλα, ας πούμε, κτλ. Ε, στη NASA κτλ. Ε, ξέρουμε ότι και τα πανεπιστήμια έχουν ανάγκη και, τα, και οι εταιρείε έχουν ανάγκη αυτές τις γυναίκες. Υπάρχει ένα κορίτσι που είπε ότι η όλη προσπάθεια στην αρχή με φόβιζε. Αλλά τελικά άλλαξα γνώμη. Είναι πολύ σημαντικό να, να, κάνουν αυτή, να περάσουν σε αυτή την διαφορετική αντίληψη κοπέλε. Επίσης, υποστήριξη προς την κοινότητα. Δηλαδή, ε, προσπαθούμε να σπάσουμε αυτή την απομόνωση, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτή την δικτύωση χάρη στα κοινωνικά μέσα σαν το Twitter, το Facebook κτλ. Ε, μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή την ομάδα ομοτήμων, ας πούμε, ε, να αντικαταστήσουμε αυτή που δεν θα υπάρξει στην τάξη ή στα, στις φοιτητικές αιστείες ή στις κοινωνικές, στη κοινωνική του ζωή στα πανεπιστήμια. Ε, μην ξεχνάτε ότι η έρευνα ε, στα πανεπιστήμια ε, έχει γυναίκες σε ποσοστό 11 με 13% μόνο. Ε, είναι πολύ σημαντικό να υποστήριξουμε νέες γυναίκες, όπως εμένα με υποστήριξαν ε, όταν ήθελα να διαλέξω μια τέτοια τεχνολογική καριέρα και να καταλάβουν ότι δεν είναι οι μόνες που ε, προσπαθούν. μιλάμε για εναν εφταετή ορίζοντα που αντιμετωπίζουν αυτές οι γυναίκες, δηλαδή ε, εξοικειώνονται με το πρόγραμμα ήδη από το γυμνάσιο, το λύκειο ε, και συνεχεία τους δίνουμε και και δάνειο, τις βοηθάμε ε, με υποτροφίες κτλ. Δημιουργούμε σχέσεις μεταξύ αυτών και των επιχειρήσεων. Οι νέες γυναίκες από το πρόγραμμά μας δηλαδή παρουσιάζονται στη ΣΥΣΚΟ, ε, στη Βόρεια Καρολίνα, ε, για να βρουν δουλειά στον τομέα της πληροφορική. το να βρούμε τις γυναίκες λοιπόν, κάνουμε την προσπάθεια ήδη από το γυμνάσιο και το λύκειο. Ε, μερικά από αυτά που πετύχαμε. Το κάνω αυτό εδώ και πέντε χρόνια. Ξεκίνησε το 2008. Έχουμε πάνω από 10.000 γυναίκες οι οποίες έχουν γραφτεί. Έχουμε 2.300 κορίτσια που συμμετείχαν σε διάφορες τελετές. 88% ε, έχουν πάει σε πανεπιστήμιο, σε τεχνολογικές και επιστημονικές ε, κατευθύνσεις. Ε, έχουμε 1.600 εθελοντές, ενήλικες και πολλούς άντρες μεταξύ αυτών. Έχουμε 50 πολιτείες που συμμετέχουν, 54 ε, ε, ομάδες που τιμούν, περιφερειακές ομάδες που τιμούν περίπου 1000 κορίτσια, δίνουν δηλαδή με έμπρακτο τρόπο, βραβεύουν 1000 κορίτσια το χρόνο. Αυτή είναι η κατάστασή μας, ε, πώς εξελιχθήκαμε μέσα σε πέντε χρόνια στις ΗΠΑ και το κόστος ανακορής ήταν κάτω από 100 δολάρια. Ε, είναι απλό αυτό που κάναμε, είναι αποτελεσματικό, χαμηλού κόστους και δεν είναι ολοκληστορία. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ε, ότι μια κοπέλα, ας πούμε, είναι καλή σε αυτό, να της το πούμε, να μπορεί να το κάνεις ε, και να της δώσουμε την υποστήριξη. Ε, Πολλοί άνθρωποι, α πούμε, κάποια στιγμή όταν κοιτάνε, πίσω τη ζωή, κοιτάνε τη ζωή τους και το παρελθόν τους, θυμούνται κάποιον που τους βοήθησε και τους ενθάρρυνε. Ε, είναι σημαντικό αυτό που κάνουμε γιατί ε, δεν μπορούμε, είναι κάτι που δεν μπορούν να το κάνουν οι καθηγητές. Έχουμε μια τεχνολογική πλατφόρμα επίση που το υποστηρίζει και ελέγχει όλα τα δεδομένα ε, και η ομάδα μου συνεργάζεται με πανεπιστημιακούς Αυτές είναι οι πληροφορίες μας, που έχω να σας δώσω και να μια φωτογραφία από τις πρώτες τις σκαπανής γυναίκες ε, στον κλάδο. Κοιτάξτε τις. Ευχαριστώ λοιπόν και την ε, Φάρμερ. Τώρα θα πρέπει να διακόψουμε τις ε, παρεμβάσεις. Έχουμε σημειώσει πλέον μια κάποια καθυστέρηση και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Σάνμπεργκ. Thank you. We have now Mrs. CEO of Facebook, joining. Είναι η διευθύνουσα σύμβουλος του Facebook, κυρία η οποία θα μας μιλήσει μέσω σύνδεσης βίντεο. Καλώς ήρθατε κυρία Σάντρα. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας τόσο νωρίς το πρωί. Σας δίνω το λόγο αμέσως. Με την ελπίδα ότι θα μπορέσετε να μείνετε μαζί μας για να απαντήσετε ενδεχομένως και σε σχόλια και ερωτήσεις από τα μέλη μας. Έχετε το λόγο κυρία Σάνμπεργκ. Πρέπει να εξηγήσω ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ακροατήριο γεμάτο κορίτσια και προσβλέπουμε ιδιαίτερα αυτά που θα μας πείτε και αυτά που θέλετε να πείτε για το μεγάλο αγώνα στον οποίο αποδιόμαστε για την μεγαλύτερη παρουσία των γυναικών στις τεχνολογίες Σας δίνω το λόγο λοιπόν. Άφωνα τα χείλη της κυρίας Σάντμπεργκ Έχουμε κάποιες δυσκολίες, θα προσπαθήσουμε και πάλι. Μάλιστα. Ήθελα οι τελευταίες σειρέ να έρθουν μπροστά, ούτω ώστε να δώσουμε μια εικόνα έτσι γεμάτη αίθουσα στην ομιλητριά μας. Σας παρακαλώ, όσοι κάθεστε πίσω, πίσω, ελάτε μπροστά, εκεί που είναι οι θέσει των Ευρωβουλευτών. Μην τρέπεστε, ελάτε. Γιατί έτσι όπως το βλέπουμε από αυτή την πλευρά, μοιάζει άδεια η αίθουσα, είναι κρίμα. Yeah, please. Yes, please. Yeah. Okay. Yeah, please take the chair. Yeah, go on. Yeah.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 Yeah. We should work on the evidence of commons and non-commons. Yeah. Yeah. Otherwise, we'll take one this way. Yeah. Yeah. Yeah. Allora proponiamo di continuare le nostre relazioni, poi quando avremo il Μπορούμε να συνεχίσουμε και τις ομιλίες και όταν έχουμε τη σύνδεση θα διακόψουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν να επανέλθετε στις θέσεις σας και θα δώσω το λόγο στην Ντόνα Μέσλα.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 Σκεφτόμαστε γιατί ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών που επιλέγουν να σπουδάσουν πληροφορική είναι τόσο ε, χαμηλός, ε, με οδήγησε σε τέσσερις συστάσεις. Αλλά θέλω να σας πω δύο λόγια για μένα, για να καταλάβατε πώς ε, οδηγήθηκα σε αυτές τις συστάσεις. Λέγομαι Ντόνα Μέσλερ και δουλεύω ως System Administrator σε ένα γραφείο στο Άμστερνταμ. Ε, μεγάλωσα στο Cape Town της Νότιας Αφρικής και ήμουνα ε, έφηβη μέσα στη δεκαετία του 80, όταν τέλειωνε η εποχή του Απαρτχάιντ. Συμμετείχα ε, στο κίνημα κατά του Απαρτχάιντ και συζητούσα πολιτική με τους ε, συμφοιτητές μου. Πήγαινα σε συναντήσεις στο χώρο της Εκκλησίας και αυτή η περίοδος με επηρέασε βαθύτατα. Επηρεάσει την προσωπικότητά μου. Νομίζω ότι έμαθα να σκέφτομαι με κριτική σκέψη, ε, με δημιουργικότητα. Ε, έμαθα να σκέφτομαι για τον εαυτό μου, αλλά μου αρέσει να συμμετέχω στην ε, κοινωνία, να εμπλέκομαι σε ό,τι συμβαίνει γύρω μου και να προσπαθώ για να βελτιωθεί ο κόσμος. Κάτι άλλο ενδιαφέρον, όταν είσαι λευκό κορίτσι στην ε, Νότια Αφρική είναι ότι είχα την ευκαιρία να φοιτήσω σε πολύ καλά σχολεία στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Ε, φυσικά, τι πρέπει να πω, κάτι το αντιφατικό εδώ. Χάρη αυτό το καθεστώ του Απαρτχάιτ, τα σχολεία, τα δημόσια σχολεία, δημοτικά και γυμνάσια, χρηματοδοτούνταν αφιδώς. Ε, σαν να ήταν δημο, ε, ιδιωτικά σχολεία. Τα δημόσια σχολεία λοιπόν ήταν καλά χρηματοδοτούμενα. Ε, επίσης οι καθηγητές μου ήταν θαυμάσιοι και φαντάζομαι ότι είναι πολύ ευχάριστο να δουλεύει κανείς σε ένα πλούσιο σχολείο. Ας πάμε τώρα στον επόμενο αιώνα. Ή μάλλον, είμαι τώρα το 2001 και μπαίνω σε ένα hack club που λέγονταν ASCII στο Άμστερνταμ. Ε, μιλάμε τώρα για ένα εργαστήρι, φανταστείτε, των υπολογιστών ε, απίστευτος χώρος μοναδικός. Ε, ήταν ε, σε ένα υπόγειο κάτω από ένα βιβλιοπωλείο, ήταν σκοτεινό, δυσάρεστο, γεμάτο από καλώδια, κομπιούτερ, ε, μόνιτορ. Ήταν σαν να βρίσκεσαι σε μία έκθεση, ας πούμε, με κολάζ και τα λοιπά. Και το πιο εντυπωσιακό ήταν ο κόσμος εκεί πέρα. Ε, είχαν την ιδέα ότι το ίντερνετ θα πρέπει να είναι ελεύθερο και για όλους. Και αυτό το έκαναν πράξη. Είχαν, πήραν το χώρο αυτό, ε, ήταν ελεύθερος ε, σε όλους, δωρεάν, και πλήρωναν την ευρυζωνική σύνδεση από την τσέπη τους. ανακύκλωναν όλο το υλικό ΙΤΑΙ και άρχισαν να έχουν και ομάδες συζητήσεις και εργαστήρια. Εγώ συμμετέχω λοιπόν σε αυτά τα εργαστήρια. Ήταν πολύ σημαντικές αυτές τις στιγμές στη ζωή μου, γιατί συνειδητοποίησα ότι πρόκειται για ένα νέο σύνορο που θα επηρεάσει την κοινωνία και τον κόσμο γύρω μου. Αποφάσισα λοιπόν να παρατήσω τη δουλειά μου ως νοσοκόμα και να βρω δουλειά στον τομέα της πληροφορικής. Ήμουν ε, ήμουνα ήδη τριαντάρα και τότε και αισθανόμουν ότι ο, τρόπος, ε, ο μόνος τρόπος για να καταλάβω τι συμβαίνει γύρω μου ήταν να βυθιστώ σε αυτό, ε, να δουλέψω σε αυτόν τον κλάδο, να είμαι κάθε μέρα ε, σε επαφή με τα κομπιούτερ. Προσπάθησα να μάθω και μόνη μου. Αυτό που κράτησα από τις μέρες στο σχολείο μου, ε, την καλή μου εκπαίδευση, είναι ότι ήμουν σε θέση να μάθω μόνη μου. Αλλά παρόλα αυτά δυσκολευόμουν με τους υπολογιστές, δυσκολευόμουν πάρα πολύ. Ε, συνάντησα και άλλες γυναίκες που και αυτές ε, ήταν, ε, ερχόταν εκεί πέρα και συχνάζαν στο άσκι. Μα τι... Και όταν ρωτούσαμε τους άντρες μια τεχνική ερώτηση στο άσκι για τα κομπιούτερς, μας, δώσαν, μας μια απόλυτα ενδελεχή, τεχνική, ευρεία, εξαντλητική απάντηση με ιδιόγλωσσα έτσι υπολογιστών, δεν καταλάβαινε τίποτα. Τίποτα. Δεν μπορούσαμε να την παρακολουθήσουμε αυτή την απάντηση αυτοί οι άντρες προέρχονταν από πολυτεχνία, ήταν μηχανική τα ύψιλον. Εμείς ερχόμασταν, είχαμε μια τελείως διαφορετική πορεία. Και εγώ ήμουν αρχάριο τόσοι ή Το ενδιαφέρον ήταν ότι όταν το συζήτησα με τις άλλες γυναίκες στο Άσκι, το θέμα αυτό, ε, συνειδητοποίησα ότι όλες είχαμε την ίδια εμπειρία. Όλες είχαμε, το βιώναμε τον ίδιο τρόπο. Αποφασίσαμε λοιπόν να βρισκόμαστε και Τώρα θα ήθελα να δείξετε τη δεύτερη μου διαφάνεια και αποφασίσαμε σε όλη την οθόνη παρακαλώ πατήστε το F. Δεν δουλεύει. Αποφασίσαμε να οργανώσουμε τη δική μας ομάδα. Να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας, ο κάθε ένας θα έπαιρνε ένα θέμα, θα το ψάχνε και θα διδάσκαμε η μία την άλλη. Ήταν σαν μια λέσχη βιβλίου, ας πούμε. Αυτή η ιστορία. Ήταν τέτοια επιτυχία που αποφασίσαμε να την ανοίξουμε αυτή την ιστορία και να δίνουμε τέτοια μαθήματα, δηλαδή να ανοίξουμε αυτό το εργαστήριο και σε άλλους. Ε, ονομάσαμε την ομάδα μας Gender Changer. Ε, ε Gender Changer είναι ένας μετασχηματιστής ουσιαστικά. Έχει ένα τμήμα με τρύπε από τη μία που είναι το θηλυκό και έχει, από την άλλη έχει τις εξοχές ε, που είναι το αρσενικό τμήμα. Ε, φυσικά δύο καλώδια, ε, μία μπρίζα ας πούμε, μα έχουμε δύο, τα σχηματιστεί με δύο τρύπε, ας πούμε, δεν, μπορεί, δεν μπορούμε να συνδέσουμε τα καλώδια πήραμε αυτό το όνομα. Το άλλο που ήταν ελκυστικό στην, στο εργαστήρι μα είναι ότι αποφασίσαμε να το ανοίξουμε μόνο σε γυναίκες. γιατί, λόγω της εμπειρίας μας. Από την ε, εμπειρία μας με τα εργαστήρια ε, είπαμε ότι, είδαμε ότι καλό είναι να έχει μια ομοιογένεια η ομάδα για να διδάσκεται καλύτερα. Εμείς ε, αντιμετωπίσαμε τότε πολύ μεγάλη αντίδραση από τους άντρες που ήταν και πλειοψηφία στο Hack Club εκεί στο Άμστερνταμ. Ε, κάναμε πάρα πολλές συζητήσεις, αλλά αποφασίσαμε να συνεχίσουμε έτσι, γυναίκες μόνο δηλαδή. Και μετά, μετά από μία εβδομάδα ε, ζητούσαμε από τους συμμετέχοντες να μας πούν τι πίστευαν για αυτή την ε, ιδέα, ότι είναι μόνο για γυναίκες. Οι περισσότερες γυναίκες ήταν θετικές απέναντι σε αυτή την ιδέα. Συνεχίσαμε λοιπόν έτσι, μόνο για γυναίκες και δεν το μετάνιωσα. Συνέχισα να δουλεύω και να οργανώνω εργαστήρια. Θα ήθελα να σας δώσω δύο παραδείγματα από εργαστήρια που οργάνωσα. Ε, νομίζω ότι είναι σημαντικές και για τις συστάσεις που θα σας πω. Καταρχάς, ε, στο Rotterdam, στο Fox University, έδωσα ένα εργαστήρι για ενήλικες. για το hardware. Ε, οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν ε, ηλικιωμένοι, ήταν το ανοιχτό πανεπιστήμιο αυτό. Ε, οι περισσότεροι ήταν ηλικιωμένοι και δεν είχαν πολύ σχέση με υπολογιστές, αλλά δεν σταματούσαν και η αξιολόγηση ήταν πολύ θετική. Ε, οποιοδήποτε περίπλοκο θέμα, αν το δώσεις, αν το διδάξεις με τον κατάλληλο τρόπο, μπορεί να το μάθει ο άλλος. Αυτό είναι το βασικό. Επίσης, ε, δεύτερο παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν, στο, σε φοιτητές ανθρωπολογίας ε, αυτό το, οργάνωσα ένα εργαστήρι για ένα εργαστήρι με το μάθημα ήταν φυσικά hardware, δηλαδή υλικό ηλεκτρονικό υπολογιστών, αλλά ήθελα κυρίω να του διδάξω την έννοια του vendor lock-in. Ε, αυτό που συνειδητοποίησα από, από το εργαστήριο αυτό είναι ότι κανένα δεν είχε δει το εσωτερικό ενό υπολογιστή από όλου αυτού του ανθρώπου. Ε, κάθε μέρα πρέπει να παίρνουμε αποφάσει ε, στη ζωή μα για την τεχνολογία. Και αν δεν καταλαβαίνουμε καθόλου αυτή την τεχνολογία, πώ θα επιλέξουμε σωστά. Αυτό είναι αυτό που κατάλαβα. Και τώρα, α πάμε στι τέσσερι συστάσει μου. Η πρώτη είναι, είναι ότι πρέπει να ψάξεις ε, παντού όταν αναζητάς συμμετέχοντες. Όχι μόνο τους νέους, αλλά και τους γέρους. Τους ε, εργαζόμενους και τους άνεργους. Και τους επιστήμονες, αλλά και τους καλλιτέχνες. Ποτέ δεν ξέρεις πού θα, που θα βρεις ανθρώπους με ενδιαφέρον. Μπορεί διάφοροι από όλους αυτούς να θέλουν να αλλάξουν καριέρα εκεί που δεν το περιμένεις. Στην ομάδα μας λοιπόν, <laughs> αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μία μόναχα από πολλές ομάδες αυτές. Η Donest στη Βαρκελόνη, μια αντίστοιχη οργάνωση στις Βρυξέλλες. Με ακούτε, με ακούτε. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες μας. Έχουμε τόσα πολλά πράγματα να κάνουμε και οργανώνουμε εργαστήρια, ατελιέ και ποτέ δεν πρόκειται να σταματήσουμε αυτές τις προσπάθειες. Η δεύτερη σύσταση που θέλω να σας δώσω Μπορώ να συνεχίσω. Ναι, είναι το να δημιουργήσετε μια σωστή στάση. Πρέπει τα κορίτσια να ξέρουν ότι είναι δυνατές, ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Το, τα ατελιέ μας δεν μας έκαναν ιδιαίτερα εξειδικευμένες προγραμματίστρες. Όλα αυτά τα οποία κάνουμε είναι γιατί αυτό το οποίο θέλαμε να κάνουμε έπρεπε να το κάνουμε πιστεύω ότι δεν είναι μοναχα το θέμα της ικανότητας, είναι η αφοσίωση, είναι η θέληση να κάνει κανείς κάτι. Η τρίτη μου σύσταση πρέπει να μαγεύονται τα νεαρά κορίτσια, να κρατάμε αυτή την αίσθηση του μαγικού που έχουμε όταν είμαστε μικροί και βλέπουμε τον ουρανό να είναι μπλε. και να μην χάσουμε αυτό από το σχολείο και τη σχολική εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε να αλλάξουμε την εικόνα της τεχνολογίας. Η τεχνολογία δεν είναι για την τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι κάτι το οποίο είναι παντού, παντού γύρω μας. Αν κάνω μια αναδρομή στη δική μου ζωή, άλλαξα καριέρα και πέρασα στην τεχνολογία, γιατί κατάλαβα ότι και ο κόσμος γύρω μου άλλαζε με ένα ραγδαίο τρόπο και ήθελα και εγώ να συμμετέχω σε αυτές τις αλλαγές. Πολλοί άνθρωποι δεν το βλέπουν έτσι. Βλέπουν τεχνολογία ως ηλεκτρονικά, gadget, υπολογιστές και κώδικα προγραμματισμού. Αν θέλουμε να προσελκύσουμε περισσότερες κοπέλες όμως, πρέπει να κάνουμε Πρέπει να, πούμε, να τους δείξουμε ότι όλα αυτά είναι παντού. Ευχαριστώ. Ζητώ αλλά δεν μπορούσαμε πάνω από 13 λεπτά. Σας ευχαριστώ για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεσή σας. Ελπίζω τώρα να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, αλλά θα πρέπει όλοι και όλες να φορέσετε τα ακουστικά σας. Cheryl, use your opportunity now for we are in. Um, honorable members of the European Parliament, uh, Chairperson Sartori and Gustavo. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Αναφέρεται στα ονόματα των μελών του Προεδρείου. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας σήμερα, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι το θέμα των νέων γυναικών στην ε, τεχνολογία της πληροφορικής είναι κάτι το πάρα πολύ κρίσιμο για όλες τις περιοχές του κόσμου και για την επιχείρησή μας. Εγώ τον τελευταίο καιρό έχω ασχοληθεί πολύ με τις γυναίκες σε, ίδιο, σε ηγετικές θέσεις, διότι είναι λίγες μέχρι τώρα. έχουν το 1 πέμπτο των θέσεων των βουλευτών σε όλο τον κόσμο, είναι το 17% των μελών των διοικητικών συμβουλίων και δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο όπου οι άνδρες να μην είναι ε, υπεύθυνοι των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων σε ποσοστό 95%. Οι φωνές των γυναικών λοιπόν δεν ακούγονται με σωστό τρόπο. Το ίδιο λοιπόν ισχύει σε όλο σχεδόν το κόσμο. 30% είναι το πολύ οι γυναίκες, για κάθε χίλιες γυναίκες με πανεπιστημιακό πτυχίο 29, 29 μόνο έχουν πτυχίο στον τομέα της πληροφορικής. Και μειώνονται οι αριθμοί αυτοί και στις Ηνωμένε Πολιτείε σήμερα. Το 1985 οι γυναίκες ήταν περίπου το 35% αυτών που έπαιρνε πτυχίο στην πληροφορική, ενώ το ποσοστό αυτό έχει πέσει στο 18%. Και η έλλειψη λοιπόν γυναικών στις ηγετικές θέσεις και η έλλειψη των γυναικών στην τεχνολογία έχει ένα τεράστιο οικονομικό κόστος στις κοινωνίες μας και στις χώρες μας. Αν δει κανείς, τη μείωση αυτή θα δει ότι δεν υπάρχουν αρκετοί για να καλύψουν τις ανάγκες. Αν υποθέσουμε ότι θα έχουμε ακριβώς το ποσοστό το ίδιο ανδρών και γυναικών, τότε στις συνεμένες Πολιτείες ε, θα καλυφθούν όλες οι ελλείψεις που υπάρχουν στο προσωπικό στην πληροφορική. Αν οι γυναίκες μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις ικανότητές τους στο ίδιο ποσοστό επαγγελματικά με τους άνδρες, τα πράγματα θα βελτιωθούν ιδιαίτερα. Κάποιος έλεγε ότι ένας από τους λόγους που η κατάσταση δεν πηγαίνει καλά είναι ότι το πεδίο δεν είναι δίκαιο για τις γυναίκες. στην ουσία ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού μένει εκτός της διαδικασίας σπουδών και ενασχόλησης με τον συγκεκριμένο χώρο. Τα στερεότυπα δυστυχώς κυριαρχούν. Κυκλοφόρησαν t-shirt στις Ηνωμένε Πολιτείε με στερεότυπα. Σε, σαν παράδειγμα οι κοπέλες φόραγαν t-shirt τα οποία έλεγαν ότι είμαι πάρα πολύ όμορφη για να ασχολούμαι με τα μαθήματά μου στο σπίτι και θα τα κάνει ο αδελφός μου που είναι καλύτερος σε αυτά από μένα. Τέτοια στερεότυπα δυστυχώς αναπαράγουν μια κατάσταση η οποία παρεμποδίζει την παρουσία των γυναικών στις σταδιοδρομίες για την τεχνολογία της πληροφορικής. αν ε, γνωρίζεις καλά τα στερεότυπα, τα ακολουθείς τελικά, είναι ένα δηλητήριο. Γιατί ως κορίτσια μας λένε ότι εμείς είμαστε για άλλα πράγματα. Και προτού κάνουμε ένα τεστ μαθηματικών ή οτιδήποτε τέτοιο, μας έχουν προειδοποιήσει ότι το φίλο μας δεν μπορεί να τα κάνει καλά. Αλλά οι κοπέλες τα καταφέρουν πολύ καλά στα τεστ αυτά, άμα δεν τους μιλήσει κανείς. Είναι τα στερεότυπα τα οποία ενισχύονται συνέχεια σε όλη μας τη ζωή. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και με την έννοια του υγείστε. Λέμε σε μια κοπέλα η οποία έχει ηγετικό ρόλο ότι προσπαθεί να κάνει το αφεντικό όταν παίζει ένα ηγετικό ρόλο. Εγώ που σε όλη μου τη ζωή δεν έχω ακούσει ποτέ να λένε σε ένα αγόρι ότι το παίζει μεγάλος και αφεντικό. Αλλά σε όλο τον κόσμο για τα κορίτσια αυτό ισχύει και γι' αυτό λέω όταν πρόκειται να πείτε αντί να πείτε σε ένα κορίτσι ότι το παίζει αφεντικό να της πείτε ότι έχει πραγματικά τις δεξιότητες ενός διευθυντή. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο δεν είναι αστείο. Αυτό όλο δεν είναι αστείο. Έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση. Ένα αγόρι που έχει ηγετικές ικανότητες, αυτό θεωρείται δεδομένο. Όταν όμως ένα κορίτσι έχει αυτές τις ίδιες ικανότητες, τότε γελάνε όλοι. Αυτό πρέπει να αλλάξει σε επίπεδο νοοτροπή, γιατί δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Πρέπει να τις ενθαρρύνουμε με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τα αγόρια. Το ίδιο ισχύει και για τις για τους εργαζόμενους. Την προηγούμενη εβδομάδα σε πόλεις, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Βερολίνο, στο Λονδίνο, έχω κάνει το ίδιο πράγμα. Είπα στο ακροτήριο, αν είστε άνδρες και σας έχουν πει ότι, σας έχουν πει ότι έχετε ηγετικές ε, ικανότητες και σας έχουν πει ότι είστε υπερβολικά, μάλλον επιθετικό στη δουλειά, σηκώστε τα χέρια. Μα κανείς δεν σηκώνει το χέρι του. Αυτά συμβαίνουν. Αν είσαστε γυναίκα και σα έχουν πει ότι είσαστε πολύ επιθετικοί στη δουλειά σα σηκώστε το χέρι σα. Όλες οι γυναίκε σηκώσαν το χέρι του. Και εκεί, όπω και εδώ. Αυτό κάνουν τα ακροατήρια παντού. Οι περισσότεροι άνδρες δεν θεωρηθούνται ποτέ επιθετικοί. Και όλες οι γυναίκες που είναι επαγγελματίες θεωρούνται ότι είναι πάρα πολύ επιθετικές. Γιατί όλα αυτά είναι τα στερεότυπα. Θεωρείτε ότι οι γυναίκε εδώ είναι πιο επιθετικές από τους άνδρες. Η έρευνα λέει ότι μάλλον οι άνδρες είναι πιο επιθετικές. Απλώς περιμένουμε όλοι τους άνδρες και τις γυναίκες να συμπεριφέρονται διαφορετικά. Όλα αυτά τα στερεότυπα είναι αυτό το οποίο εμποδίζει τις γυναίκες να μπουν στην τεχνολογία. Περιμένουμε τα γόρια μας να γίνουν προγραμματιστές, να είναι καλοί στις επιστήμες, τις θετικές και τα μαθηματικά και λέμε στα κορίτσια με άμεσους και με έμεσους τρόπους ότι δεν περιμένουμε κάτι αντίστοιχο από αυτές. Και προστατεύουμε πάρα πολύ τα παιδιά μας από το διαδίκτυο. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά σε όλο τον κόσμο οι γονείς προστατεύουν πάρα πολύ τα κορίτσια τους από ότι τα αγόρια τους. Αφήνουμε τα αγόρια μας να ψάχνουν και να διερευνούν και τα κορίτσια τα προσέχουμε πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν τα κορίτσια δεν μπαίνουν στην πληροφορική, δεν τα ενθαρρύνουμε. Λέμε στους γονείς λοιπόν αφήστε τα κορίτσια σας στην τεχνολογία. Αφήστε τα και μην προσπαθείτε να τα εμποδίσετε. Δεν είναι καλύτερα λοιπόν τα πράγματα αυτή τη στιγμή πέρσι το καλοκαίρι. Η κόρη μου που ήταν 7, ο γιος μου 7 χρονών πήγε στο Πανεπιστήμιο του Στένφορντ σε ένα θερινό πανεπιστήμιο για πληροφορική. Αυτοί που αποφασίζουν σε αυτήν την ηλικία είναι οι γονείς. Πήγε λοιπόν σε αυτά τα μαθήματα. Και Μόνο δύο κορίτσια ήταν εκεί, η ανιψιά μου και μια φίλη της. Όλα τα άλλα παιδιά στο μάθημα πληροφορικής ήταν αγόρια. Και κάτι αντίστοιχο γίνεται στις δικές σας χώρες. 35 αγόρια και δύο κορίτσια μοναχα ή πέντε κορίτσια στην πραγματικότητα. Δεν βελτιώνονται λοιπόν τα πράγματα. Και όταν σου λέω για τα προγράμματα που έχουν σε άλλα μέρη του κόσμου, όλα αυτά τα προγράμματα είναι γεμάτα αγόρια και καθόλου κορίτσια. Μο, όταν λοιπόν οι κοπέλες φτάσουν στο πανεπιστήμιο, ήδη υπολείπονται. Και δεν παίρνουν πια μαθήματα πληροφορικής, γιατί νιώθουν ότι υστερούν. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κορίτσια μας, να του πούμε ότι είναι καλές στα μαθηματικά και στις θετικές επιστήμες, στις χώρες στην ε, Ασία, που γίνεται κάτι τέτοιο, τα κορίτσια τα καταφέρουν καλύτερα από τα αγόρια. Σχεδόν σε όλους τους τομείς. Στη Γαλλία οι κοπέλες είναι 64% των πανεπιστημιακών πτυχίων στο πρώτο επίπεδο. Αν πούμε λοιπόν ότι αν πούμε στα κορίτσια ότι θα είναι καλά, θα μπορέσουν να τα καταφέρουν. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα παιδιά μας θα έχουν πρόσβαση, ίση πρόσβαση στις τεχνολογίες. Πρέπει να παίζουν video games, να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές, να χρησιμοποιούν τεχνολογία και να μην τις εμποδίζουμε. Και κυρίως πρέπει να αλλάξουμε τα στερεότυπά μας για τις γυναίκες και τα κορίτσια, γιατί μονάχα αλλάζοντα αυτά τα στερεότυπα θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα για τις τεχνολογίες ICT και τα προβλήματα αυτά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για το χρόνο σας και θα είμαι έτοιμη να απαντήσω σε ερωτήματα ενδεχομένω. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις. Η Επίτροπος καταρχήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας αφιερώνεις και για την έμπνευση που μας δίνεις. Εσύ επισκέφθηκε στην Ευρώπη πριν από λίγο, από ό,τι ξέρω, για να παρουσιάσεις την προσπάθειά σου. Ούτως ή άλλως ε, πολλοί από εμάς ξέρουμε, ξέρουμε το εγχείρημά σου. Υπήρχε διαφορετική αντίδραση εδώ στην Ευρώπη από ό,τι στην Αμερική. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Υπάρχουν σημαντικές πολιτιστικές διαφορές μεταξύ όλων των χωρών και προφανώς μεταξύ των ΗΠΑ ε, και των επιμέρους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αλλά ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια και μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ Ασίας και ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής το βιβλίο μου έχει δημοσιευθεί σε 24 χώρες και σε κάθε χώρα έχω μια ειδική ομάδα με που δουλεύει για τη συγκεκριμένη χώρα με τις ε, τοπικές στατιστικές και την τοπική έρευνα. Και κοιτάξτε, σε όλε τις ε, χώρες πολύ περισσότεροι άντρες ασχολούνται από ότι γυναίκες ε, και τα αγόρια χειροκροτούνται γιατί ασχολούνται, ενώ τα κορίτσια τα κρατάμε. Δεν τους δίνουμε τις ευκαιρίες. Ούτως ή άλλως περισσότερες χώρες τα κορίτσια τα πηγαίνουν το ίδιο καλά με τα γόρια και μερικές φορές και καλύτερα. Ας πούμε στη Γερμανία 51% κορίτσια, στη Γαλλία 64% και σε μερικές χώρες παραπάνω. Ξέρουμε ότι τα κορίτσια μπορούν να μάθουν, να ηγηθούν, αλλά ξέρουμε επίσης ότι δεν τα ενθαρρύνουμε αρκετά. Επίσης δεν ενθαρρύνουμε τα κορίτσια αρκετά να κατευθυνθούν προς επιστημονικές κατευθύνσεις. Πρέπει να καταλάβουμε τα μοντέλα και για κάθε χώρα και για τον πλανήτη ολόκληρο. Ε, Ευχαριστώ. Η συνάδελφος κυρία Χέρτσογκ. Χαίρομαι που στο χώρο της πληροφορικής μπορούμε να σας συναντήσουμε. Συζητάμε σήμερα το απόγευμα Όταν οι άνδρες επιλέγουν δεν θα είναι οι γυναίκες, ε, δεν πρέπει να είναι οι γυναίκες ε, η καλύτερη επιλογή. Όπως ακριβώς γίνεται και σε μία σχέση γάμου. Σε αυτή τη φάση οι άνδρες κυριαρχούν τον κόσμο της πληροφορικής. Πώς μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να γίνουμε αυτό που είπα πριν, η επιλογή τους. Ταυτόχρονα όχι μόνο οι άνδρες κυριαρχούν στον χώρο της πληροφορικής, αλλά δεν είναι και η καλύτερη περίπτωση. Εννοείται πως οι γυναίκες όχι. Πως ο κόσμος που κυριαρχείται από τους άνδρες ε, δεν γίνεται από τις γυναίκες δεκτό. Λοιπόν, πως θα κάνουμε λοιπόν τις γυναίκες την καλύτερη επιλογή, αυτό κατάλαβα. It's amazing to get through that and stay in that. Κοιτάξτε, το θέμα είναι να προσπαθήσει κανείς να είναι ενεργός. Οι γυναίκες έχουν πάρα πολύ ταλέντο, αυτές οι γυναίκες. Και όσο προχωράμε στην προσπάθεια που κάνουμε, τόσο θα χάνονται τα στερεότυπα. Η απάντηση που δίνουν πολλοί άνδρες είναι δεν τους αρέσει η πληροφορική γιατί δεν τους αρέσει η πληροφορική. Ενώ οι άνδρες πηγαίνουν επειδή υποτίθεται τους αρέσει. Δεν είναι φυσικά αυτή η ισχυρισμή σωστή. Βλέπουμε ότι οι γυναίκες μπορεί να έχουν ηγετικές δυνατότητες. Αλλά πρέπει να τις δούμε πρώτα για να αρχίσουμε να συνδέουμε τις γυναίκες με τις ηγετικές δυνατότητες. Και οι γυναίκες που είναι στον χώρο σήμερα θα ανοίξουν το δρόμο για μας εμείς θα ανοίξουμε την πόρτα για να μπουν στο χώρο μας οι επόμενες γυναίκες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συζητήσατε μαζί μας σήμερα. Χαιρετίσματα στην Καλιφόρνια. Σας ευχαριστώ. Bene, collegamento ε. Ωραία. Σταματάει εδώ η σύνδεση και μπορούμε τώρα να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας μετά από αυτή την σύνδεση και τη συνομιλία με μια γυναίκα που έχει τόσο σημαντικό ρόλο, τόσο σημαντική θέση γιατί το Facebook μπήκε στη ζωή όλων μας, μπορούμε να κλείσουμε αυτή τη μέρα. Αλλά πριν κλείσουμε θα δώσω το λόγο στην Ίντι Ταντών, που είναι η κύρια εμπειρογνώμονας και εκπαιδεύτρια μιας ε, ομάδας. Δεν είπατε τη σωστή ομάδα, τη διορθώνει η ενδιαφερόμενη, την πρόεδρο. I'm sorry, but they have the wrong PowerPoint on. Uh, good afternoon, my name... Είναι από το ITU. Ε, λέγομαι Νίδη. είμαι α, από την α, Νότιο Αφρική. Ε, εδώ και πολλά χρόνια, περίπου 22 χρόνια είμαι εκπαιδεύτρια, περίπου τη μισή μου ζωή δουλεύω με τις γυναίκες στην Αφρική, στην Καραϊβική, ε, κεντρική Ευρώπη και κεντρική Ασία και προσπαθώ να εντάξω την πληροφορική στην ζωή τους και να προσαρμόσω την, ε, πληροφορική για τις ανάγκες τους. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. είναι τιμή να είμαι εδώ σε αυτήν την αίθουσα με τόσες πρωταθλήτριες της αλλαγής. Η, η ITU ε, μου ζήτησε να κάνω μια παγκόσμια αξιολόγηση για τις δεξιότητες που θα χρειαστούν ε, στο χώρο της πληροφορικής στο μέλλον και τι πρέπει να γίνει, ούτω ώστε οι γυναίκες και τα κορίτσια α, θα έρθουν σε επαφή με αυτόν τον αναπτυσσόμενο τομέα. Ακούσατε πάρα πολλά για όλο το απόγευμα γι' αυτό, δεν θα τα επαναλάβω, αλλά κοιτάξτε, αυτή η έκθεση που σας δείχνω είναι online και οι συναδελφοί μου από το ITU ε, έχουν μια μεγάλη βαλίτσα με φυλάδια τέτοια ε, στα αγγλικά και γαλλικά και ε, άλλες γλώσσες, αλλά όχι σουαχίλι. Το βιβλίο έχει πάρα πολλές στατιστικές. Φερρυπίν. Στις χώρες του ΟΣΑ οι, γυναί... γυναίκες συμμετέχουν πολύ λιγότερο στον τομέα της πληροφορικής και όμως ε, το μερίδια τους ε, στην απασχόληση συνολικά αυξάνεται. Στην Εστονία και Ουγγαρία που είναι πάνω από το μέσο όρο του ΩΣΑ, οι γυναίκες ε, είναι το 45%. Αλλά σε εξειδικευμένες καριέρες, στις ΗΠΑ έχουμε 25%, εν συνεχεία Ισλανδία, Φιλανδία και Ουγγαρία έχω την αίσθηση ότι ακούσατε ένα κάρο στατιστικές και έχετε μπουχτήσει για σήμερα. Ε, να σας πω και το τελευταίο από στατιστικές. Όπως είπε και κάποιος συνάδελφος, η ITU έχει φτιάξει και ένα, τη δικτυακή πύλη παράλληλα με αυτό το φυλάδιο και έχει και πρακτική πληροφορία ε, για τις γυναίκες και τα παιδιά που θέλουν να αποκτήσουν ε, μια καριέρα σε αυτό το τομέα. Μπορείτε λοιπόν να επισκεφθείτε τον ιστοτοπό μας από την 1η ε, Ιανουαρίου του 2013 μέχρι στιγμής. Είχαμε 20.000 επισκέψεις στην δικτυακή πύλη. Το 75% ήταν καινούργιοι. Είχαμε παλιούς αλλά και καινούργιους. Ε, όταν ξεκίνησε το ITU είχαμε 220 προγράμματα, ε, τώρα έχουμε 526. Ε, έχουμε δυνατότητα για επιχορηγήσεις, μαθητείες, στάζ και τα λοιπά. Οι συναδελφοί μου ενθαρρύνουν τα κορίτσια και τα αγόρια όμως να μπουν σε αυτό το κλάδο. Και οι εταιρείε, οι οργανώσεις ε, και οι κυβερνήσεις έχουν προγράμματα που υποστηρίζουν γυναίκες. Ε, θα ήθελα αυτή την ε, πληροφορία να την επικαιροποιείτε και να επεκτείνετε τους πόρου που υπάρχουν. Τι μπορώ να πω εγώ που δεν ακούστηκε σήμερα. Θα ήθελα να εστιάσω σε δύο θέματα που συνδέονται. Μια στιγμή. Το, θέμα το, το ένα θέμα είναι το πώς. Πώς θα φτάσουμε στα κορίτσια και θα τα κρατήσουμε στον τομέα και το δεύτερο, πού θα τα ψάξουμε, πού είναι αυτές οι γυναίκες και πού είναι οι θέσει αυτές του μέλλοντος. Για να σας ετοιμάσω για τις απαντήσεις μου σε αυτά τα ερωτήματα, θα σας πω... Θα σας μιλήσω για κάποιες γυναίκες σε αυτόν τον κλάδο, έτσι, τυχαία. Και λόγω του, της προέλευσής μου, έτσι, θα σας δείξω καταρχήν τρεις γυναίκες από ε, επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις. Ε, το όνομά τους δεν είναι σημαντικό, η εταιρεία τους, το όνομα της εταιρεία δεν είναι σημαντικό, αλλά το τι κάνουν είναι σημαντικό. Αυτή, ας πούμε, η κοπέλα είναι, προσπαθεί να ε, ε δει, ας πούμε, το νερό ε, ε, υγεία λοιπά, Πώς μπορούν να, αυτές οι υπηρεσίες να παρασχεθούν με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Δεύτερον, ε, πάλι για τις υποδομές. Τι λέει αυτή η γυναίκα. Ε, με αυτόν τον τρόπο και να το μούμε, όλα όσα νομίζαμε ότι ξέραμε για ένα σύστημα, τα πήραμε και τα πετάξαμε και μάθαμε ε, εκ νέου. Ε, και το σύστημα για το οποίο μιλάει είναι υποδομές νερού σε μια πόλη. Ε, με τα SMS μπορούν 18.000 χρήστες να δουν που υπάρχει η πλησιέστερη πηγή νερού στην κατοικία τους. Ε, μια άλλη εδώ λέει ότι η επόμενη πρόκληση τα επόμενα 50 χρόνια πιστεύω θα είναι να δημιουργήσουμε αξιοπρεπή εργασία για όλους. Όχι η ελεημοσύνη, αλλά μέσω των δυνάμεων της αγοράς. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει ένα σύστημα πληροφορικής και δίνει απλές θέσεις ε, σε ανθρώπους ε, που ήταν αποκλεισμένοι από τον κλάδο αυτό, όχι μόνο στην Ινδία, όχι σε Ινδούς δηλαδή, αλλά και σε ανθρώπους από την ΑΕΤ και τα λοιπά. Μιλάμε για κοινωνικές επιχειρηματίες. Κοιτάξτε το ήθος που έχουν και η διοντολογία που έχουν. Υπάρχουν άλλες δύο γυναίκες, μία ε, είναι ηγέτης σε μία κλασική επιχείρηση πληροφορικής, είναι ε, Κινέζα, ε, είναι, έχει συνειδρήσει μία εταιρεία ημιαγωγών και η άλλη δεν έχω την εικόνα της, αλλά λέγεται η εταιρεία της Mashery και είναι μια, εφαρμογή, μια πλατφόρμα εφαρμογής ε, Α, εσεί ε, γνέφετε, α, άρα καταλαβαίνετε περί τίνο πρόκειται. Ε, η Intel ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει τη Mastery. Τι σα λέει αυτό? Οι γυναίκε μπορεί να ηγούνται σε κάποιες παραδοσιακές μορφές ICT, αλλά βρίσκονται στην εχμή του δόρατος σε πολλές εφαρμογές που έχουν να κάνουν με δίκτυα. Και το τελευταίο παράδειγμα είναι η κυρία Σερ Βάγκα, η οποία ίδρυσε την HTC. Πρέπει, μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες. Πάρα πολλές αυτές οι γυναίκες κάνουν αυτούς τους οργανισμούς για φιλανθρωπικούς ε, λόγους. Βοήθησε χιλιάδες να αποκτήσουν αυτές τις ε, ταμπλέτες HTC και η ελπίδα της είναι ότι οι γυναίκες αυτές θα μπορέσουν ε, να δημιουργήσουν ένα πιο ενεργό ρόλο για αυτές και για εκατομμύρια ακόμα ανθρώπων θα μπορέσουν να ακολουθήσουν τον δρόμο μεγαλύτερη ευμάρειας στο μέλλον. Πιστεύω ότι οι γυναίκες πρέπει να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στη τεχνολογία, όχι μόνο ως χρήστες, αλλά και ως ε, πηγές καινοτομία, ως επικεφαλής επιχειρήσεων και επικεφαλής του βιομηχανικού αυτού κλάδου. Τι μας λέει λοιπόν αυτά τα πορτρέτα. Όταν κάνουμε λοιπόν τη μελέτη μας, να είναι συνεχιστές στην επόμενη διαφάνεια. Θα πω πράγματα που είπανε και οι συναδελφοί μου, ότι τα αγόρια προτιμούν όλα αυτά τα θέματα γιατί έχουν να κάνουν με βιντεοπαιχνίδια κτλ. Και οι γυναίκες δεν ασχολούνται. Αλλά όταν τα κορίτσια καταλαβαίνουν ότι η ICT μπορεί να τους δώσει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν καλύτερα και να αλλάξουν τον κόσμο, τότε πραγματικά αλλάζει τα πάντα. Είτε είναι θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης ή θέματα περιβάλλοντος ή αν είναι να φροντίζουν τη γιαγιά τους, δεν έχει σημασία. Υπάρχει αυτή η πτυχή του να αλλάξει κανείς τα πράγματα στον κόσμο και νομίζω ότι αυτό προσελκύει τις γυναίκες Ας συνεχίσουμε λοιπόν αυτή την ε, στάση. Χρειαζόμαστε επομένω και την ε, επίσημη εκπαίδευση, τα κέρια τα θέματα. Χρειαζόμαστε να υπάρχει και κάποια δυνατότητα να λειτουργούν κάποιες αμέντορες και να βοηθούν την εκπαίδευση και επίσης πρέπει να προετοιμαστούμε για νέες οικονομικές δραστηριότητες, νέες μορφές, γιατί θέλουμε να μεταφέρουμε στην επόμενη γενιά την θέληση να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα που έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε τεράστια πίεση, έχουμε ε, ανισότητες οι οποίες ε, αυξάνονται συνέχεια, το όπως καταδεικνύει και από τους ε, συντελεστές Gini που φτάνουν δυσθεωρητά ύψη. Επομένως, θα πρέπει να συνεχίσω και να πω πού είναι οι γυναίκε. Υπάρχει ο δείκτης για το τρίτο δισεκατομμύριο και λέει ότι ένα δισεκατομμύριο γυναίκες θα μπορούσαν να μπουν στην οικονομία στην επόμενη δεκαετία ως ε, εργοδότε, ως εργαζόμενες και ως στελέχη επιχειρήσεων. 865 εκατομμύρια γυναίκες θα είναι σε ηλικία εργασίας 20 με 65 μέχρι το 2020 και θα έχουν δυνατότητα να συμβάλλουν στην εθνική του οικονομία. Από αυτές σε 865 εκατομμύρια γυναίκε, 812 εκατομμύρια είναι σε αναδυόμενε και αναπτυσσόμενες χώρες. Και ήμουν σε ένα συνέδριο που μιλούσε για το, το συνέδριο για το πού θα βρούμε τον επόμενο Bill Gates ή Steve Jobs. Μάλλον γιατί ο επόμενος Bill Gates Steve Jobs θα είναι γυναίκα και θα γεννηθεί σε μια αναδυόμενη χώρα. Σύντομα συμπεράσματα. θα σας υπενθυμίσω τρεις α, ε, συνομιλίες, γιατί μου αρέσουν περισσότερο αφήγησεις. Η πρώτη είναι από μια γυναίκα η οποία είναι σε μια εταιρεία software στο, από το Πανεπιστήμιο Κιαμπόγο και την ξέρω πολύ καλά αυτή την εταιρεία και μου είπε στο τηλέφωνο δεν ασχολήθηκα με το, την πληροφορική για τις επιχειρήσεις αλλά πήγα στο Κιαμπόγο Πανεπιστήμιο που είναι ένα μικρό πανεπιστήμιο κάνοντας ε, πληροφορική και το διάλεξα αυτό γιατί η τεχνολογία εξακολουθεί να προχωράει, να αλλάζει κάθε μέρα και ήθελα πραγματικά να διερευνήσω περισσότερο τις τεχνολογίες. Όπως είπε και η συνάδελφος από την Νότια Αφρική, ήμασταν περίπου 20 κορίτσια και 80 αγόρια. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτή η μαθητεία θα με βοηθήσει να βρω δουλειά σε κάποια εταιρεία. Η δεύτερη αφήγηση είναι από τις ΗΠΑ, από μια γυναίκα η οποία ασχολείται με τη στελέχωση στις ΗΠΑ για τα θέματα της πληροφορικής. Και για πρώτη φορά λέει, καταλαβαίνουν αυτές οι γυναίκες που ασχολούνται με τη στελέχωση πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουν να προσελκύσουν τις γυναίκες, οι οποίες είναι πολλές φορές πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Συνήθως δεν θεωρούν ότι μπορούν να επιτύχουν δεν νομίζω ότι μπορούν να επιτύχουν, αλλά εγώ νομίζω ότι μπορούν να συμβάλλουν πάρα πολύ. Όταν μιλώ με μία γυναίκα που βρίσκεται σε αθητεία, μου είπε πως το σχέδιο για το γονιδίωμα είχε 200 οι οποίοι ήταν όλοι άντρες και όταν ζήτησαν μόνο γυναίκες για ένα αντίστοιχο πρόγραμμα πήραν 100 αιτήσει για τρεις θέσεις μονάχα. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε να υπάρχει καλύτερο software με το να μην εμποδίζουμε τις γυναίκες να συμμετέχουν γιατί είναι καλύτερες ε, συγγραφείς λογισμικού. Τέλος, μια συνομιλία με ένα ε, στέλεχος μιας εταιρείας που τώρα ξεκινάει για το Web 2.0. Είπε ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούν πολύ περισσότερα την κοινωνική διαδικτύωση από τους άνδρες. Αυτές κυριαρχούν στον κοινωνικό ε, κυβερνόχωρο. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν γιατί η οικονομία, το αναψώμενο κομμάτι της οικονομίας βρίσκεται εκεί. Μπορεί μετά από τρεις μήνες ε, εκπαίδευσης μια γυναίκα να, δι, να σχεδιάζει καλύτερες ε, εφαρμογές από τους άντρες, γιατί είναι πιο διαισθητικές και έχουν μια πιο ανθρωπιστική προσέγγιση. Σέριλ Μίλλερ είπε το πρωί ότι πρέπει να στοχεύσουμε ψηλά. Αυτό είναι το απαραίτητο. Θα πρέπει αυτό το ψηφιακό στόχος μας να πάει πάρα πολύ ψηλά. Το θέμα δεν είναι οικονομικό μόνο, αλλά είναι το θέμα της υγείας και της οικολογίας για το μέλλον μας. Ευχαριστώ. Όπως είδατε έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας για λόγους επιμελητίας θα δώσω το λόγο για να κλείσει η Επίτροπος τη συνάντησή μας. Έχετε το λόγο, κυρία Κρούς. Να σας ευχαριστήσω εγκάρδια και εσάς την ίδια προσωπικά σαν πρόεδρο της Ήτρε, να ευχαριστήσω την Εντίθ Χέρτσοκ και τις συναδέλφους της για τις πρωτοβουλίες σας. Είμαι βέβαιη ότι αυτά που λέω εκφράζουν όλους που συμμετέχουν εδώ. Θα ήθελα να κάνουμε μια συμφωνία όλοι μαζί. Αν συμφωνούμε όλοι για αυτά τα οποία ακούστηκαν από τις διάφορες ομιλήτριες και από τη Σέβιλ Σάνμπεργκ, να ξεφορτωθούμε τα στερεότυπα. Θα πρέπει όλες αυτές οι στατιστικές να αποδείξουμε ότι πάνε λάθος. δεν αυξάνεται είναι αλήθεια ο αριθμός της εμπλοκής των γυναικών στην πληροφορική, αυτό είναι σαφές, αλλά θα το αλλάξουμε αυτό. Γιατί διαπιστώνουμε ότι είναι λάθος η κατεύθυνση αυτή και θα στοχεύσουμε ακόμα ψηλότερα. Αυτό θα αλλάξει τα πράγματα στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν ας κάνουμε μια συμφωνία. Εσείς θα επιστρέψετε στα σπίτια σας, θα μιλήσετε με τους φίλους σας, συνεργάτες σας, τα παιδιά σας. Και να πείτε δεν θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα αποδεχθούμε την κατάσταση αυτή. Δεν θα αποδεχθούμε τα στερεότυπα. Τότε μόνο θα αλλάξουν τα πράγματα. <clears throat> γιατί πιστεύουμε στην, στον σχεδιασμό των ρόλων που καλούμε να αναλάβουμε και τα πρότυπα δεν θα πρέπει να αφορούν μόνο τις διάφορες σέριλ. Τα πρότυπα είστε εσείς, τα πρότυπα είναι οι γειτόνισές σας, τα πρότυπα είναι όλων οι γείτονε και οι γειτόνισες, αρκεί να αποδείξουν ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και έτσι θα προχωρήσει ο κόσμος. Πρέπει να αλλάξουμε την κοινωνία αυτό έχει μεγάλη σημασία. Μία από τις ομιλήτριες είπε ότι χάρη στο θάρρος της άλλαξε τη ζωή της. Μπορούμε να εμπνευστούμε όλοι μας ότι αν ακολουθήσουμε την εύκολη, την ασφαλή οδό, δεν θα βγούμε κενδυσμένοι. Όχι κενδυσμένοι. Ε, ποια είναι τα πρότυπα, εσείς είστε τα πρότυπα. Εξηγήστε σε όλους τους φίλους σας ότι όλοι μπορεί να είναι πρότυπα. Έτσι αλλάζουν οι νοοτροπίες. Και τελευταίο, ευχαριστώ όλους σας, την Πρόεδρο, την Εντίτ. Ε, εμείς είμαστε στην υπηρεσία σας ας παραμείνουμε σταθεροί. Εάν ε, επιμείνουμε θα βρούμε λύση. Ας βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Ας ε, δώσουμε τα χέρια γυναίκες και κορίτσια. Ας αλληλοβοηθηθούμε. Σας ευχαριστώ. Καταπληκτική δουλειά κάνατε. Ευχαριστώ την Επίτροπο, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ τους εισηγητές. Και η κυρία Χέντζοκ τελευταία. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να, θράτω, να, να αδραχθώ τις ευκαιρίες για να πω ότι αυτή ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να περάσουμε το σημερινό απόγευμα. Ελπίζω για την επόμενη ακρόαση, την επόμενη συνδιάσκεψη, θα μπορέσουμε να κάνουμε θα την κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι σε όλη την Ευρώπη θα μπορούν να παρακολουθούν τι λέμε, να μπορέσει να περάσει το μήνυμα ότι δεν είμαστε μονάχα η καλύτερη επιλογή αλλά ότι είναι σημαντικός και από οικονομική έποψη ο ρόλος των γυναικών. Μία τεχνική ανακοίνωση μετά από την συνάντηση θα υπάρξει μία δεξίωση αλλά πρέπει να πάμε στο ισόγειο, στο σαλόνι των βουλευτών για να πάρουμε ένα ποτήρι κρασί στην ρεσεψιόν αυτή. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.